Okay. Everybody, you've had, you've had a few minutes to settle down. Ναι, καθίστε παρακαλώ λίγο, Πρόεδρος. Thank you. Can, can you. can you all sit down, please, because we... Καθίστε αν θέλετε, γιατί είναι ε, φορτωμένη η ημερήσια διατάξη και έχουμε πολλές ψηφοφορίες. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε, λοιπόν. Περνάμε στο 10 της ημερήσιας διάταξης για τους ε, διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων στην εξέταση των τροπολογιών. Αντιλαμβάνομαι ότι οι μεταφράσεις ε, των τροπολογιών κατέφτασαν πολύ καθυστερημένες, ωστόσο ο εισηγητής θεωρεί ότι μπορεί να υπάρξει και να γίνει μια πρώτη χρήσιμη ενταλλαγή απόψεων γιατί έχει προγραμματιστεί και για τις 16 Μαρτίου μια δεύτερη ανταλλαγή απόψεων. Να δώσω λοιπόν το λόγο στον εισηγητή για να μας παρουσιάσει το θέμα. Ζαν Πολ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, δύο μικρές ανακοινώσεις πρώτα απ' όλα. Ένα λεπτό κατά ανώτατο όριο θα για κάθε τροπολογία. Δεύτερον, ζητώ συγγνώμη από τους πρασίνους τους φίλους μας γιατί σίγουρα χαλάσανε δάση ολόκληρα για να υποβάλουν τέτοιες τροπολογίες. Ελπίζω να μην μου το προσάψουν την ώρα της ψηφοφορίας. Καλά κάνατε επίσης και η ε, Πρόεδρε και είπατε ότι αργοπόρησαν οι τροπολογίες, δεν φταίνε οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου. Ε, 1669 υπήρχαν, αφήστε που ήταν και περίπλοκες, οπότε οι υπηρεσίες ε, κατέρευσαν κάτω από το βάρος των τροπολογιών Πάντως, είναι πολύ χρήσιμο να γίνει η πρώτη εξέτασή τους. Ο κάθε βουλευτής γνωρίζει τις δικές του τροπολογίες και άρα θα τις υποστηρίξει. Και επίσης, θα σας ενημερώσω για τις διάφορες ε, επαφές που έκανε, προκατακτικές ε, επαφές. Πολλαπλές επαφές, έτσι, τις μέτρησα. 110 ε, συνδιαλέξεις με τους εκπροσώπους των ομάδων ειδικών συμφερόντων, τους λομπίστες όπως τους λέμε και εμπλουτίστηκαν έτσι οι γνώσεις μου, αλλά δεν χρωστάω και τίποτα σε κανέναν. Επίσης ε, συζήτησα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προφανώς με την Ισπανική Προεδρία που ανέλαβε μετά τη Σουηδική. Στο Στρασβούργο έκανα κατηδίαν με όλους τους κοιόδης και με όλους τους συναδέλφους ε, που θέλησαν να με δουν ε, παρότι είναι προκατακτικές οι διατυπώσεις που επιλέξαμε και θα επανέλθουμε. Λοιπόν, για το χρονοδιάγραμμα. Σήμερα θα γίνει ανταλλαγή απόψεων. Θα ρίξουμε περισσότερο φως στην υπόθεση. Τις 16 Μαρτίου θα τα ξαναπούμε. και είναι λίγο φιλόδοξο, αλλά ελπίζω ότι στις 16 θα έχω στη διάθεσή μου τις συμβαστικές τροπολογίες που τώρα συζητούνται. Θα ρίξουμε ακόμη περισσότερο φως λοιπόν σε όλα τα θέματα και στις 12 Απριλίου όπως έχει προβλεφθεί νομίζω θα μπορέσει να γίνει ψηφοφορία και θα συζητήσουμε βέβαια με τους συναδέλφους, την Ισπανική Προεδρία, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συμμορφωθούμε με το προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα και να επιτελέσουμε το στόχο μας, να είναι αποτελεσματικό, ρεαλιστικό το κείμενό μας και να μην καθυστερήσουμε πολύ. Γιατί αν αργήσουμε υπερβολικά και δεν υλοποιηθούν οι απαιτούμενες νομοθετικές πράξεις, ε, αυξάνουμε τους κινδύνους για το μέλλον. Λοιπόν, μετά από όλε αυτέ τι συζητήσει που έκανα με του συναδέλφου επαγγελματίε, του Σκιώδη, την ε, Προεδρία, την Επιτροπή, ε, είμαι σχετικά αισιόδοξο. Έχουμε καλέ πιθανότητε να καταλήξουμε σε ένα ε, συμβαστικό κείμενο. Α μην προτρέχουμε όμω έτσι και πρέπει να παραμείνουμε ρεαλιστέ. Αλλά έχουμε καλέ πιθανότητε. Ε, σε αυτούς τους 4 πεντε μήνες ε, σημειώθηκαν ε, εξελίξεις ε, στις απόψεις των ΜΕΝ και των ΔΕ. Οι επαγγελματίες αντιτίθεντος σε οποιοδήποτε ρύθμιση. Δηλαδή, συμφωνούμε με την οδηγία, αλλά τελικά πρέπει να αφαιρέσουμε πολλά στοιχεία. Αλλά ξέρετε, άλλαξαν γνώμη, εν πάση περιπτώσει δεν ήταν τόσο απόλυτη οι επαγγελματίε αντιλαμβάνονται, όπω είπε και ο Επίτροπο στην ακρόασή του, ότι στον χρηματοπιστωτικό τομέα χρειάζεται ρύθμιση, χρειάζεται εποπτεία. Αυτή λοιπόν η θετική στάση μας επέτρεψε να κάνουμε ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων για αμυγός τεχνικά ζητήματα, ούτως ώστε η ε, εκπονηθήσα νομοθεσία να επιτελεί το στόχο της. Ποιος είναι αυτός? Να αποφύγουμε τους συστημικούς κινδύνους και να μην ε, επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας ε, στις χρηματοπιστωτικές αγοράς. Ε, δεν ρυθμίζουμε επειδή μας αρέσει να εκπονούμε νέες νομοθεσίες. Ο στόχος είναι να έχουμε αποτελεσματική και ρεαλιστική νομοθεσία η οποία λαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα του, της χρηματοπιστωτικής βιομηχανίας. Οπότε το πεδίο πρέπει να είναι ευρύ, όπως το ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ό,τι δεν είναι ΟΣΕΚΑ, ό,τι δεν είναι αλλακτικά, ε, ό,τι δεν ε, είναι οργανισμός συλλογικών επενδύσεων πρέπει να καλυφθεί από αυτή την οδηγία. Πρέπει να καλύψουμε μικρά, ε, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να καλύψουμε ειδικευμένα ταμεία ή μικρά ταμεία και γι' αυτό προτείνω δύο διαφορετικές ε, μεθοδολο, ε, μεθοδολογίες. Πρώτον οι ορισμοί. Τι δεν συνιστά ταμείο. Πρέπει να το ορίσουμε για να μην υπάρξουν ψευδεστήσει ή αδικαιολόγητοι φόβοι είναι ένα holding ε, ε, βιομηχανικής συμμετοχής ε, εξορισμού δεν είναι ταμείο εκτός και αν ο στόχος είναι να είναι ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων. Τι ούτω τρόπος πρέπει να έχουμε μια αναλογικότητα. Δηλαδή, η αναλογικότητα πρέπει να είναι ουσιαστική, να μην μείνει μόνο στη θεωρία και να ισχύουν ομοιόμορφοι κανόνες για όλους. Και γι' αυτό προτείνω, έχοντα διαβάσει ε, όλες τις τροπολογίες, ε, προτείνω να ορίσουμε τους κανόνες της αναλογικότητας και μάλιστα να πούμε ότι κάποια εγχώρια ταμεία, εγχώρια κεφάλαια που ήδη ρυθμίζονται με ικανοποιητικό τρόπο να μεριμνήσουμε ώστε να ε, συμμορφούνται και με τις απαιτήσει τη οδηγία και να μην χρειαστούν περαιτέρω διατυπώσεις ε, για αυτά τα κεφάλαια. Ε, τώρα, εάν υπάρχει ένας μόνο επενδυτής, που... ένας επαγγελματίας που χρησιμοποιεί αυτά τα επενδυτικά κεφάλαια για τις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητές του, ε, σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται οι διαχειριστές αυτών των κεφαλαίων να έχουν επιπρόσθετες απαιτήσει πληροφορίας εφόσον έχουν ένα μόνο επενδύτη. Δεν μπορεί να υπάγονται στους ίδιους κανόνες σαν να υπήρχαν πολλαπλοί επενδυτές. Ε, κατόπιν, ε, με τις παρατηρήσεις των συναδέλφων ε, τροποποίησα και εγώ ελαφρώ τη θέση μου και σας είπα ότι ούτως ή άλλως ούτω η άλλω ηταν βαση εργασία η αρχικη μου θέση σε σχέση με τις ε, τρίτες χώρες, ε, σε αυτό αναφέρομαι. Ε, θα πω και αυτό και μετά θα ακούσω τους συναδέλφους, διότι κατά τα λοιπά ακολουθώ την γραμμή που μοιάζει πολύ με αυτή που σας είχα εκθέσει την πρώτη φορά. Ε, δεν θέλουμε ε, να είναι οχυρό η Ευρώπη, αλλά ούτε και κόσκινο. Ε, είχα υιοθετήσει μια συντηρητική θέση γιατί δεν είχα βρει άλλη λύση και μου φαίνεται λίγο ουτοπική θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, έχοντας ακούσει όλους τους συναδέλφους, ε, σήμερα τελικά αποφάσισα να προτείνω ένα διαφορετικό σύστημα με δύο περιόδους, μια μεταβατική περίοδο, ε, τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια, εμείς θα το αποφασίσουμε αυτό, κατόπιν μια ύστερη περίοδο. Κατά τη μεταβατική περίοδο ε, θα συνεχίσουν να ισχύουν οι εθνικοί κανόνε για του επενδύσει ε, και τα κεφάλαια των οποίων οι επενδυτέ είναι εκτό Ευρώπη θα συνεχίσουν να θέτουν σε εμπορία τα προϊόντα του, όπω σήμερα. Κατά τη διάρκεια αυτή τη μεταβατική περίοδου ε, θα προσπαθούμε να βρούμε την ισοδυναμία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι εποπτικέ αρχέ τη χρηματοπιστωτική αγορά. Μετά την πάροδο αυτή τη περίοδου, μετά από 3-4-5 χρόνια, θα πρέπει να βρούμε μία λύση γνωρίσουμε την ισοδυναμία ε, για την ε, τάδε χώρα που βρίσκεται ο επενδυτή εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και άρα ο διαχειριστή θα εξομοιωθεί με τον διαχειριστή τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δύναται να θέτει σε εμπορία ε, τα προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχει το διαβατήριο του, του, του κεφαλαίου. Εάν δεν κατοχυρωθεί η ισοδυναμία, η θέση σε εμπορία των προϊόντων θα απαγορευτεί μετά τη μεταβατική περίοδο απολύτω μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έχουμε μία ρήτρα grandfathering διατήρηση του κεκτημένου, τόσο ώστε τα ε, κεφάλαια που θα υπάρχουν στην ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ η οδηγία θα συνεχίσουν να υφίστανται ούτω ώστε να μην υπάρξει βίαιη ρήξη ε, για κάποιε δραστηριότητε. Αυτά για τι τρίτε χώρε. Αυτό είναι ο προσανατολισμό τη νέα μου πρόταση και ελπίζω οι συζητήσεις που θα κάνουμε τώρα να μας ε, βοηθήσουν να διαπιστώσουμε αν η πρόταση αυτή συμμορφώνεται με ε, τις επιθυμίες όλων ή αν χρειάζεται επανεπεξεργασία. Αυτά, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ήθελα να σας εκθέσω αυτά τα στοιχεία. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Δεν τις διάβασα ακόμη όλες τις 1670 τροπολογίες, αλλά υπόσχομαι ότι θα το κάνω και θα ακολουθήσω τις προτάσεις των συναδέλφων Σκιωδών και άλλων και θα τα ξανασυζητήσουμε. Ελπίζω οι συναντήσεις μας ε, να γίνουν ε, μετά ε, την 5η, 6η Μαρτίου, γιατί τότε θα έχω καταλήξει στις πρώτες συμβαστικές τροπολογίες. Ανάμεσα στις 5 και 6 Μαρτίου και τις 16 θα έχουμε λοιπόν επαφές και ελπίζω να καταλήξουμε σε συμβιβασμό και θα ήθελα να σας δείσω και μια χάρη, Πρόεδρε. Ε, μπορείτε να δώσετε το λόγο στο Wolf Klintz μετά από μένα γιατί οπωσδήποτε πρέπει να φύγει, έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις ε, και τον περιμένω με ανυπομονησία να δω τι έχει να πει. Ευχαριστώ. Ε, right. Ah. Ναι, έχετε το λόγο, λέει η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντως, βιάζομαι ιδιαίτερα. Γι' αυτό σας ευχαριστώ για την εξαίρεση που μου κάνατε για να μου δώσετε το λόγο από τους σοσιαλδημοκράτες. Φαίνεται ότι έχουν προχωρήσει λίγο τα πράγματα. Δεν συνδέεται το τώρα του κόσμου με, το, με την οδηγία αυτή μιλάμε για τους συστημικούς κινδύνους ε, και αναφέρεται ότι θα δημιουργηθούν τέτοιοι κίνδυνοι. Ελπίζω ότι οι διαβουλεύσεις μας να έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο προκειμένου να έχουν αντισκεδαστεί πλέον αυτοί οι φόβοι. Έχουμε μία σειρά τροπολογιών, την οποία υποβάλαμε. Θα τις δείξω εν συντομία. Ιδάλλως δεν θα είχαμε χρόνο καθόλου. Καταρχάς ζήτησα οι όροι όπως μας υποβλήθηκαν να επιστραφούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ζητήσουμε να αντικατασταθούν από δύο οδηγίες, μία για τα hedge funds και μία για τα private equities. Ξέρω ωστόσο ότι τέτοια δυνατότητα, τέτοια πιθανότητα μάλλον είναι πολύ περιορισμένη. Ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εκπροσωπείται και από τον νέο Επίτροπο Μπαρνιέ τα βλέπει πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Θέλει να καλύψει όλα τα ταμεία, όλες τις επενδύσεις. Παρ' όλα αυτά ε, θεωρώ ότι τα hedge funds και τα private equities είναι αυτά τα οποία ε, είχαμε ως στόχο και θα έπρεπε να έχουμε ως στόχο. Κατά δεύτερον, το πεδίο εφαρμογής. Οι Στου οποίου αναφέρεται η οδηγία αυτή. Όπω είπε ο Πολ, υπάρχει μια σειρά τέτοιων ταμείων. Δεν είναι μόνο αυτά που ανέφερε, τα ειδικά ταμεία στην ε, Γερμανία, είναι και τα investment grants στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία είναι σίγμανα στο χρηματιστήριο, τα family trust στην Σουηδία και το καθεξής. Και ανέφερε ο εισηγητή ότι αυτά μπορεί να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή της οδηγίας, αλλά από τη στιγμή που ρυθμίζονται επαρκώ εθνικά, θα πρέπει να θεωρούνται ως ισότιμοι αυτή η ρύθμιση και δεν χρειάζεται ε, να επιβληθούν νέα γραφειοκρατικά τέτοια εμπόδια. Έκανα μία πρόταση ανέφερα ως ποσό για τα leverage funds τα 500 εκατομμύρια. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα α, απελευθερωθούν από κάθε όρο. Υπόκειται άλλωστε στην οδηγία αυτή, ωστόσο θα πρέπει να πληρούν τις ε, όρους διαφάνειας. Αυτό σίγουρα θα οδηγήσει σε κάποια ελάφρυνση. Σε ό,τι αφορά το evaluation, την αξιολόγηση, το είπα και με την λογική αυτή που και της τροπολογίας μας, ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει ε, αξιολόγηση τρίτου μέρους. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε απλά ότι η αξιολόγηση θα γίνεται από ανεξάρτητες αρχές και αυτή η ανεξαρτησία μπορεί να γίνεται, να εγγυάται αν θέλετε και ο έλεγχος να γίνεται από ένα τμήμα της επιχείρησης. Η ευθύνη τώρα για την αξιολόγηση και τα αποτελέσματά της είναι στον ε, manager των Alternative Investment Funds, των ε, εναλλακτικών επενδύσεων. Γιατί στην περίπτωση που υπάρχει τρίτος αξιολόγητης, η ευθύνη είναι δικιά του. Θεωρώ επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, μία ρύθμιση αποθεματικής τράπεζας και θα πρέπει να διατηρηθεί αυτή η ρύθμιση. Και όρισα τα καθήκοντα. Ποια είναι τα καθήκοντα της τράπεζας αυτής. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά τις λεπτομέρειες θα πρέπει να περιμένουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα θίξει οριζόντια το θέμα αυτό. και ελπίζω πριν από την ψηφοφορία στην Ολομέλεια να συζητήσουμε τα θέματα ευθύνη. Πέμπτον, το θέμα του leverage, της μόφλευσης. Θα θυμάστε ότι στην τελευταία συζήτηση θεωρούσα ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να τεθούν συγκεκριμένε ε, απαιτήσει. Και πρέπει να ομολογήσω ότι και ο ορισμός καν του leverage, της μόχλευσης είναι πάρα πολύ δύσκολος, πιο δύσκολος από ό,τι φαίνεται εκ πρώτης ε, άποψης. Γι' αυτό λοιπόν θα συμφωνήσω με τις προτάσεις ε, του Συμβουλίου, αλλά αποδέχομαι επίσης ότι τα κράτη-μέλη σίγουρα μπορούν να επιβάλλουν διατάξεις, όρους. Δεν συμφωνώ με τον Ζαν Πολ, με τον εισηγητή, που λέει ότι το ίδιο το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να μπορεί να καθορίσει την ε, μόχλευση. Τα κράτη-μέλη ίσως. Έκτον, τα asset stripping. Αυτό μπορεί να αφορά τα private equity αλλά και τα hedge funds ενδεχομένω. Θεωρώ ότι στο σημείο αυτό κάτι πρέπει να γίνει. Γιατί αν μπορεί να μην αποτελούν την ε, πλειοψηφία, την πλειονότητα των περιπτώσεων, οι περιπτώσεις αυτές του asset stripping, αλλά υπάρχουν. Όποιο συμμετέχει λοιπόν σε μία επιχείρηση με σκοπό, με την ελπίδα να πετύχει μία τέτοια προστιθέμενη αξία, και αυτό συμβαίνει στις, στα private equities, θα πρέπει να αφήσει τουλάχιστον τρία έτη τις μετοχές του στην εταιρεία αυτή και όχι να περιμένει σε χρόνο ρεκόρ τέτοια κέρδη σε ό,τι αφορά τώρα κατά έβδομον την τρίτη χώρα. Όπως είπε και ο Ζαν Πολ, συμφωνώ που θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα καταστεί ούτε οχυρό ούτε φυλακή. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε συμφέρον να υπάρχει εισρωή κεφαλαίου προς την Ένωση και Θα πρέπει να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα εφιστάμενα καθεστώτα. Ε, εγώ είμαι υπέρ των 5 ετών, τώρα δεν έχω όμως κάποιος, ε, κάποια προτίμηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει τα στα επόμενα 5 χρόνια θεωρώ να προσπαθήσει να βρει ε, ισότιμες συμφωνίες. Και αν το καταφέρουμε αυτό, όντως θα μπορέσουμε να δώσουμε ένα τέτοιο διαβατήριο, αν θέλετε, σε αυτές τις ε, επιχειρήσεις των τρίτων χωρών. Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προσπαθήσει να συντονίσει όσο γίνεται τα 27 καθεστώτα και αν δεν συμβεί αυτό το οποίο δυστυχώ είναι και πιθανό να αναπτύξει μετά από 5 χρόνια ένα 28ο καθεστώ ευρωπαϊκό. Αυτά λοιπόν προς το παρόν και ελπίζω από τις προηγούμενες συζητήσεις με τον Ζαν Πολ και από τις άλλες συζητήσεις να μπορέσουμε πλέον να πούμε ε, ρεαλιστικά ότι τα πράγματα φαίνονται να είναι πολύ πιο αισιόδοξα σήμερα από ότι πριν από δύο μήνες. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ρόμπερτ, θέλεις το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ήρθα λίγο αργότερα και δεν άκουσα τον φίλο μου τον Σαν Πολ Γκοζές και ζητώ συγγνώμη ορισμένα σχόλια εντάχει. Καταρχήν, έχουμε 1669 τροπολογίες, εξαιρετικό πακέτο. Δεν είχα ούτε χρόνο ούτε διάθεση να τις ε, διαβάσω, αλλά πολλοί που συμμετέχουν σε λόμπι διατυπώνουν συστάσεις έχω έναν ικανό κατάλογο επιτάπητος. Καταγράφω λοιπόν όλες αυτές τις προτάσεις από τα λόμπι. Για μένα θα είναι αρνητικός αυτός ο κατάλογος, δηλαδή οι τροπολογίες ε, για τις οποίες τουλάχιστον εγώ δεν θα υπερψηφίσω. Εδώ έχουμε πολλά λόμπι. Θέλουμε να αρέσουμε στα λόμπι, στον καταναλωτή, σε πολλά μέτωπα. Θέλουμε μια οδηγία που μία διαποντός εξαλείφει αυτή την καλπάζουσα κερδοσκοπία που διακατέχει τις αγορές, που έχει μικρο- και μακροοικονομικές συνέπειες. Είμαι υπέρ λοιπόν μιας οδηγίας στεγανοποιημένης. Γι' αυτό θα ήθελα να ακολουθήσω τον εισηγητή μας, ιδιαίτερα όταν λέει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις. Ο συνάδελφος Κλίνς θέλει δύο οδηγίες από ό,τι κατάλαβα. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ καλή η ιδέα Βεβαίως υπάρχουν, υπάρχουν και τα private equities και τα hedge funds, τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου. Αλλά είμαι υπέρ ενός μέσου και αυτό που έχει ε, σημασία είναι να δούμε πώς ε, δρούν όλοι έτσι ώστε να υπάρχουν ίσοι όροι πρόσβασης. Πιστεύω ότι φυσικά δεν είναι οχυρό η Ευρώπη και ούτε θέλουμε να κατασκευάσουμε ένα οχυρό. Όμως θα πρέπει να δώσουμε πλεονεκτήματα σε αυτούς που βρίσκονται εντός Ευρώπης και όχι εκτός. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα κοσκίνισμα και πολλοί επενδυτές θέλουν ποιότητα, θέλουν ασφάλεια. Ε, άκουσα τη λέξη flight to quality. Εάν θέλουμε να φτάσουμε σε μια σωστή ποιότητα και σωστή εποπτεία θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο εσωτερικό μηχανισμό για τα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε να κάνουμε με μια μακροχρόνια συζήτηση που δεν είναι εύκολη. Εμείς ως σοσιαλιστές είμαστε στη διάθεση του εισηγητή για να φτάσουμε σε σωστούς συμβιβασμούς και είμαι σίγουρος ότι με το Ζαν Πολ Γκοζές θα φτάσουμε σε αυτούς του συμβιβασμού. Εάν οι πράσινοι, οι φιλελεύθεροι και άλλοι θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, είμαστε ανοιχτοί. Δεν θέλουμε όμως συμβιβασμό για το συμβιβασμό. Θέλουμε κάτι το σταθερό, το συμπαγές και να μην έχουμε αυτές τις σκανδαλώδεις πρακτικές που είδαμε τα τελευταία χρόνια. Εδώ μιλώ για τις τάσεις υπερβολικής μόχλευσης. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να ορίσουμε αυτές, αυτές τις υπερβολικές μοχλεύσεις, όμως αυτό μπορεί να συζητηθεί και νομίζω χρειάζονται σαφείς κανόνες. Αυτό ισχύει και για άλλες πρακτικές, όπως το asset stripping που απασχόλησε τον φίλο μου τον Κλίνς. Νομίζω και αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρξει ένα συγκερασμός έτσι ώστε να μην είναι τίποτα βλαβερό. το, όσον αφορά το naked short selling, δηλαδή τις ομές ανοιχτές πωλήσει, αυτό είναι ανήθικο και δεν θέλουμε να επηρεάζουμε τις αγορές. Όλοι γνωρίζουμε ότι σε επίπεδο διεθνών τραπεζών, ιδιαίτερα ε, σε επίπεδο Lehman Brothers, φτάσανε στα όρια του, της πτώχευσης εξαιτίας των ανοιχτών πωλήσεων. Εμείς θέλουμε να αφήσουμε, να εξαλείψουμε αυτή την πρακτική. Νομίζω θα πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό το ζήτημα, το οποίο θα μας συνοδέψει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Thank you. I can't see the green... Δεν υπάρχει ο σκιώδης των πρασίνων. Ποιος θέλει να μιλήσει. Ο κ. Σουάνγκίγκολτ. Πασκάλ. Δυστυχώς δεν μπορεί να παραβρεθεί σήμερα. Καταρχάς να ευχαριστήσουμε πολύ τον Σαν Πολ για τον όγκο δουλειά, δουλειάς που επιτέλεσε. Δεν ξέρω αν είχατε υποπτευθεί από πριν ότι θα λαμβάνατε τόσες πολλές τροπολογίες. Σας εύχομαι να το δισκεδάσετε και πολλές άγρυπνες νύχτες με όλη την υπόλοιπη δουλειά που σας μένει. Και εγώ έχω την εντύπωση ότι οι τροπολογίες δεν έχουν προταθεί από λομπιίστες μόνο, αλλά επειδή έχουν γραφτεί από άλλους φορείς Ουσιαστικά αυτό μειώνει την, ε, τον όγκο δουλειά, γιατί όταν τα κείμενα είναι ταυτόσιμα ουσιαστικά, δεν χρειάζεται να τα διαβάσουμε όλα και να τα αποφασίσουμε όλα. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω όλα όσα υπόθηκαν. Θα ήθελα να εστιάσω σε κάποια σημεία τα οποία θεωρώ ότι θα πρέπει να συζητηθούν εδώ στην Επιτροπή μας. Το πρώτο αφορά το βασικό θέμα του κατά πόσο η μόχλευση θα πρέπει να ρυθμίζεται ή όχι και σε ποιο βαθμό. Στο σημείο αυτό, δυστυχώς, ως τώρα βλέπουμε ότι είναι πολύ διαφορετικές και διστάμενε οι απόψεις. Καταρχάς, υπάρχει η άποψη που αποτυπώνεται στις τροπολογίες των φιλελευθέρων, οι οποίοι λένε ότι ουσιαστικά δεν θέλουμε να αναμειχθούμε στο θέμα αυτό, δεν θέλουμε να περιορίσουμε καθόλου τη μόχλευση. Και στη δική σας ε, έκθεση, κύριε Κοζές, περιλαμβάνονται μόνο λίγες και όχι πολύ ουσιαστικές ρυθμίσεις. Θεωρούμε ότι το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα συνολικά έχει υπερβολικά μεγάλη μόχλευση. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ρύθμιση. Εδώ φαίνεται ότι δίστανται όπως και παλιά οι απόψεις μας. Και εδώ πέρα παραπέμπω στο θέμα της ε, ακρόας της Επιτροπής ε, Αντιμετώπισης της Κρίσης, όπου συζητάμε τέτοια θέματα και η ομάδα μας θεωρεί σαφέστατα ότι υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα. Είναι υπερβολικά μεγάλη η μόχλευση και θα πρέπει την οδηγία αυτή να τη χρησιμοποιήσουμε για τον περιορισμό της μόχλευσης. Και το ίδιο θέμα τίθεται και σε ό,τι αφορά το τραπεζικό τομέα. Θα πρέπει να διευκρινιστεί. Και το ίδιο θεωρούμε, ήδη διαφορά ουσιαστικά υπάρχει διάσταση απόψεων, υπάρχει σε ό,τι αφορά το πώς φανταζόμαστε πόσο ενιαία θα είναι η ευρωπαϊκή αγορά σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις. Εξακολουθούν λοιπόν να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις στο σημείο αυτό. Και έχουμε και διαφορές για το ρόλο των ε, υφιστάμενων private placement regimes στο μέλλον. οι φιλελεύθεροι και οι Στριτικοί συμφωνούν ότι τα, οι επενδύσεις οι οποίες ε, ρυθμίζονται απ' έξω θα πρέπει να παραμείνουν ε, σε ισχύ σε ό,τι αφορά τα εθνικά συστήματα private placements. Είπατε, κύριε Γκοζές, ότι ε, η άποψή σας έχει αλλάξει όμως και ότι έχετε μετακινηθεί λίγο πιο πολύ προς τη δική μας κατεύθυνση. Θεωρούμε ότι δεν έχει νόημα σε μια τέτοια αγορά να μην υπάρχουν ε, ενιαίες ρυθμίσεις. Αν μάθαμε κάτι από την κρίση είναι ότι όποιος έχει τα πιο χαμηλά κριτήρια εγκατάστασης δεν ανήκει στην ενιαία αγορά. Ότι χρειαζόμαστε μία σαφή διάκριση μεταξύ της ενιαίας υποπτικής αρχής αφενός, των ενιαίων κανόνων και του ανοιχτού ανταγωνισμού στο πλαίσιο της αγοράς. Δεν θέλουμε τον κατακριματισμό των διαφόρων ε, συστημάτων εποπτείας. Ένα άλλο θέμα το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα είναι οι κερδοσκοπικές επιθέσεις στην Ελλάδα. και αυτό το θέμα καταδεικνύει με πάσα σαφήνεια την ανάγκη σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις και τις δραστηριότητε ε, να υπάρξει όντως δραστηριότητα. Ενεργοποίηση. Η κυρία Λαγκάρτ είπε σε μία σημαντική συνέντευξη ότι οι δραστηριότητες των επενδύσεων αυτών θα πρέπει να ρυθμιστούν. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε κερδοσκοπικές επιθέσεις κατά την ακυρεότητα του συστήματος του ευρώ να επιτραπούν ότι στην Ελλάδα υπάρχουν προβλήματα και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα κράτη-μέλη δεν ε, δραστηριοποιήθηκαν ενεργά για να προλάβουν τα προβλήματα αυτά, ισχύει, είναι αληθές. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπήρξαν συστηματικές κερδοσκοπικές επιθέσεις, τις οποίες επιτρέψαμε. Αυτό όμω τι σημαίνει, σημαίνει ότι η οδηγία αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί, να αξιοποιηθεί όχι μόνο για τη ρύθμιση των επενδύσεων, αλλά στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και η κερδοσκοπία σε ό,τι αφορά προϊόντα. Αυτό δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση του εισηγητή και νομίζω ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε το θέμα αυτό. Στο σημείο όπου γίνεται κερδοσκοπική ε, δραστηριότητα με τον ενεργητικό εταιριών, να, έχει, να υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης. Να μην λέμε δηλαδή ότι «Α, εντάξει, δεν πειράζει». Δεν είμαστε κατά των επενδύσεων, των εξωτερικών επενδύσεων, ασφαλώς και όχι, αλλά θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εποπτείας. Να αυτό, προβλέπεται αυτό από τη ρύθμιση και το παράδειγμα της Ελλάδας καταδεικνύει στο σημείο αυτό την ανάγκη να προχωρήσουμε παραπέρα από την πρόταση του εισηγητή. Θα ήθελα επίσης να πω ότι σε ορισμένες περιπτώσεις υποστηρίζουμε και τις τροπολογίες των σοσιαλιστών και εμείς κινούμαστε προς ανάλογη κατεύθυνση σε ό,τι αφορά το short selling, τις ακάλυπτες πωλήσει και σε ό,τι αφορά το asset stripping Νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι συζητήσεις προκειμένου να προχωρήσει παραπέρα στο σημείο αυτό η οδηγία. για να προστατεύσουμε τις επιχειρήσεις από τις πρακτικές αυτές. Και ξέρουμε φυσικό, φυσικά δεν είναι εύκολο να ορίσουμε ε, το asset stripping και πότε υπάρχει asset stripping. Αλλά έχουμε προτάσεις βάσει των οποίων μπορούμε να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας δεν θα πρέπει να πούμε ότι α, εντάξει, θα αφήσουμε τα πράγματα ως έχουν. Δεν θα ήθελα να είμαστε στη θέση σας ε, με τις 1600 πόσες ε, τροπολογίες, αλλά ελπίζουμε με τον τρόπο αυτό που ακολουθήσαμε ως τώρα να συνεχίσουμε τη δουλειά μας προκειμένου να γεμίσουμε, να πληρώσουμε τα κενά τα οποία υπάρχουν, να γεφυρώσουμε τις ε, διαστάσεις των απόψεων που υπάρχουν, ακολουθώντας την αρχή ότι μετά την κρίση αυτή κανένας φορέας δεν επιτρέπεται να μείνει χωρίς ρύθμιση. Χρειαζόμαστε εποπτεία χωρίς να πνίξουμε τις επενδύσεις, αλλά είναι σαφές ότι οι πρακτικές οι οποίες συνέβαλαν στην κρίση οι οποίες είχαν αρνητικό αντίκτυπο δεν επιτρέπεται να συνεχιστούν σε ό,τι αφορά κερδοσκοπία κατά νομισμάτων, ε, υπερβολική αφαίρεση ε, αξιών από επιχειρήσεις, υπερβολική μόχλευση. Όλα αυτά θα πρέπει να επιληθούν και θεωρώ ότι το πνεύμα που διακατέχει όλη την Επιτροπή είναι το σωστό και χαιρόμαστε και ανυπομονούμε για την περαιτέρω συνεργασία μαζί σας αγαπητέ κύριε Σιγητά. Ευχαριστώ Σαντ. Και εγώ θα ήθελα να τονίσω την εξαιρετική εργασία του κυρίου Γκοζές και το γεγονός ότι είναι ιδιαίτερα συνεργάσιμος. Θα ήθελα να περιοριστώ σε ορισμένα σημεία, διότι έχουμε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που μας απασχολεί, αλλά θα ήθελα να σας πω από πού προέρχονται οι δικές μου τροπολογίες. Είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Γκοζέ στο πρώτο θέμα και συμφωνώ με τον φιλελεύθερο σκιώδη είναι ότι θα πρέπει να μας απασχολήσουν οι καταναλωτές, η προστασία τους. Για ποιους καταναλωτές μιλάμε. Μιλάμε για τους αποταμιευτές, για τους αυριανούς συνταξιούχους και εκείνους οι οποίοι έκαναν επενδύσεις σε επιχειρηματικά κεφάλαια υψηλού κινδύνου. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούν να, μπορούν να γίνουν επενδύσεις σε ταμεία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει νομίζω να έχουμε ε, μειώσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε, μια καλύτερη, σε ένα καλύτερο συνταξιοδοτικό, έτσι ώστε να μην υπάρχουν περικοπές στο συνταξιοδοτικό όπως υπάρχουν σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δέχομαι την άποψη του κυρίου Γκοζές για τα, τη διατήρηση και εκτιμένων, grandfathering, για μια μεταβατική περίοδο γιατί είναι σαφές, θα πρέπει να είναι σαφές για άλλες δικαιοδοτικές αρχές το τι ακριβώς πρέπει να κάνουν και τι κριτήρια να ακολουθήσουν για να ε, υπάρχει ισομέρεια. Ισοβάθμιση δηλαδή, γιατί πολλές δικαιοδοτικές αρχές εκπρόσωποι τους μου είπαν ότι θέλουν να υπάρχει μια επάρκεια, μια ισοβάθμιση, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν τι σημαίνει επαρκώς αυτό και να μην το αφήσουμε για πέντε χρόνια και μετά να πούμε «Α, δεν ε, πληρούνται αυτά τα κριτήρια». Θα πρέπει να υπάρχει μια επάρκεια ήδη από τώρα. Επίσης, όσον αφορά την εμβέλεια, πρότεινα ορισμένες εξαιρέσεις γιατί θα πρέπει έχουμε ένα σαφή ορισμό αναλογικότητας. Όλοι θέλουμε την αναλογικότητα, διότι δεν θέλουμε τα μικρά ταμεία να μην μπορούν να ανταγωνιστούν τα μεγάλα. Θα πρέπει να είμαστε σαφείς τι σημαίνει αναλογικότητα. Θα ήθελα να το δούμε με τον εισηγητή και με τους σκιώδεις, έτσι ώστε να έχουμε έναν σωστό ορισμό αναλογικότητας. Όπως είπε και ο εκπρόσωπος των Πρασίνων, θέλουμε έναν σωστό ορισμό μόχλευσης, της ε, μόχλευσης. Υπάρχουν πολύ ε, εύλογα χρηματοπιστωτικά μέσα. Τα είδαμε ιδιαίτερα σε σχέση κάλυψης χρεών, αλλά θα πρέπει να μην υπάρχει ε, κακός χειρισμός των ισολογισμών. Σε σχέση με αυτή την οδηγία θα πρέπει να είμαστε σαφείς, διότι δεν μπορεί να ισχύει ένα είδος μόχλευσης για όλα τα ταμεία και για όλα τα στοιχεία ενεργητικού. Ποιος ε, έχει περισσότερη πείρα για να διατυπώσει το όλο ζήτημα θα πρέπει να δούμε τους εθνικούς ρυθμιστές για να δούμε ποια είναι τα συστήματα εθνικής αντιστάθμισης κινδύνου, αλλά και η Επιτροπή θα πρέπει να μας πει ποια είναι τα όρια των εθνικών ρυθμιστών στη ρύθμιση της ε, μόχλευσης. Αυτό αφορά την ΕΣΜΑ και άλλες αρμόδιες αρχές. Και ελπίζω να συμφωνείτε με αυτό. Εκεί αποβλέπουμε με τις τροπολογίες σε σχέση με τη ρύθμιση της μόχλευσης. Η μόχλευση δεν μπορεί να ειδωθεί μεμονωμένα σε σχέση με τα διάφορα προφίλ κινδύνου. Ένα δύσκολο ζήτημα βεβαίως είναι οι αμοιβέ. Όλοι ανησυχούμε για τις αμοιβέ, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τους ε, κανόνες του τραπεζικού τομέα, γιατί αυτοί που διαχειρίζονται τα μία, τα ταμεία ε, δεν έχουν τις ίδιες αμοιβέ και τα μπόνους εξαρτώνται από την απόδοση σε αυτό το τομέα. Και αυτό έχει σχέση με τους ίδιους επενδυτές. Ελπίζω λοιπόν να, δίνει, να γίνει μια συζήτηση για τις αμοιβέ να λάβουμε τις αρχές του T20 και του Διοικητικού Συμβουλίου Σταθερότητας, διότι οι τραπεζίτες έχουν διαφορετικές αμοιβέ από τον τομέα των επιχειρηματικών κεφαλαίων υψηλού κινδύνου. Το AIFM δεν μπορεί να διέπεται από το ίδιο καθεστώς. Δεν υπάρχει αιτιολογία. Το feed μπορεί να καλύψει και τον τομέα των ε, υπηρεσιών και δεν χρειάζεται να σταθούμε αλλού να αρκεστούμε αλλού σε σχέση με τις ρήτρε διασφάλισης. Θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση, όπως είπε ο κύριος Γκοζές, θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση τη στιγμή που πρόκειται για ένα αυτόνομο εγχείρημα. Σε σχέση με τις ακάλυπτες πωλήσει, short selling, υπάρχουν διαφορετικοί τύποι ε, ακάλυπτων πωλήσεων γιατί υπάρχουν οι οψιών και υπάρχουν οι ακάλυπτες καθεαυτές. Έχουμε, θα γίνει μια συζήτηση αργότερα. Αλλά νομίζω ότι οι ακάλυπτες ε, πωλήσει μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υπάρχει ε, ρευστότητα, αλλά ως προς τις οψιών θα πρέπει να είμαστε ε, σαφείς, δηλαδή ότι καλύπτουμε μόνο το νόμιμο σκέλος των ακάλυπτων πωλήσεων. Ως προς τη χρήση του όρου χρηματοπιστωτικά μέσα, financial instruments, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι τι εννοούμε. Σε σχέση με τους ε, αποταμιευτές μπορούν να λαμβάνουν τα ε, πιστοποιητικά που θέλουν, αλλά αυτό που έχουν σημασία είναι τα book entries που γίνονται για τους ισολογισμούς. Και αυτό που έχει σημασία είναι οι αποδόσεις, διότι η έννοια των αποδόσεων δεν έχει καμία σχέση με το book entry securities, δηλαδή με τα χρεόγραφα που καταγράφονται. Σε σχέση με την παγκόσμια εποπτεία, παγκόσμια εποπτεία σημαίνει ότι υπάρχουν ε, περιπτώσεις όπου ο θεματοφύλακας ορίζει τρίτους ως εγγυητές, κάτι το οποίο δεν προαπαιτείται. Και ο θεματοφύλακας, ας πούμε, δεν έχει μία προτίμηση σε... για μία χώρα και πρέπει να ορίσει έναν τριτεγγυητή. Θα πρέπει να υπάρχει αυτή η αρχή και όχι μόνο εκεί που προαπαιτείται νομικά. Μπορεί ε, δηλαδή να διοριστεί αλλά σε πολλές χώρες μπορεί να υπάρχουν λιγότερες επενδύσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τις αναδιόμενες οικονομίες. Δηλαδή, μπορεί να υπάρξει έλλειψη επενδύσεων στις αναδιόμενες οικονομίες ε, τρίτων χωρών. Έχω και άλλα σημεία που θα ήθελα να αναφέρω, αλλά δεν θέλω να κοιμηθείτε. Γι' αυτό θα ήθελα να συνεργαστούμε ε, μελλοντικά στο ίδιο πνεύμα που μας ε, διέπει μέχρι τώρα. Κύριε Κλούτ θέλετε και εσείς να μας πείτε κάτι από πλευράς Γκουε, γιατί είστε ο Σκιώδης. Μάλιστα, θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια. Ακούσαμε ότι δεν πρέπει να υπάρξουν εξαιρέσεις και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα, σε διάφορες τροπολογίες Ανέφερα ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την συνήθη νομοθετική διαδικασία κατά την σύσταση των ε, επενδυτικών κεφαλαίων και αυτό είναι σημαντικό για μας. Κάτι άλλο που ακούσαμε σήμερα το πρωί ε, σχετικά με τα κεφάλαια private equities. Ε, συμφωνώ με τους προλαλήσαντες. Δεν θέλω να επαναλάβω τα ίδια σχόλια. Ευχαριστώ. Η Μάρτεν Ντρες ε, μας ενημέρωσε ότι θέλει να μιλήσει όταν καταφθάσει, αλλά δεν τη βλέπω. Έχουμε 10 ομιλητές στον κατάλογο. Προτείνω χρόνο αγόρευσης 3 λεπτά, παρακαλώ. Πω την προϋπόθεση ότι δεν θα δηλώσουν κι άλλη συμμετοχή. Διαβάζω τον κατάλογο. Ε, Lulling, Ford, Bullman, και η Ντρέσεν αν καταθέσει και εγώ ίδια. Η κυρία Τζούρι θέλει να μιλήσει. Κάποιος άλλος παρακαλώ. Όχι. Ξαναλέω τρία λεπτά έκαστος παρακαλώ. Και μετά πρέπει να δώσουμε και λίγα λεπτά και στο Ζαμπόλ για να κλείσει τη συζήτηση. Γκούναρ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ τον Ζαν Πολ για τις προσπάθειες και τις ε, ικανότητες που έχει στον τομέα, το κατέδειξε και όλοι εντυπωσιαστήκαν που δήλωσε θα διαβάσει όλες τις τροπολογίες. Και πάλι εντυπωσιαστήκαμε από όλα όσα έχει κάνει από την αρχή ε, του ζητήματος. Χαιρόμαστε που το έχει αναλάβει το θέμα. Το σημαντικό είναι ότι θα κατοχυρώσουμε δυναμισμό στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Αλλιώ δεν θα έχουμε επενδύσει και δεν θα έχουμε και θέσει απασχόληση που χρειαζόμαστε για να έχουμε την χρηματοπιστωτική σταθερότητα μακροπρόθεσμα. Γιατί το λέω αυτό. Διότι ε, αυτά είναι τα συμπεράσματα όταν θέλουμε να ρυθμίσουμε το θέμα των συστημικών ε, κινδύνων. Δεν είμαι σίγουρος ότι ακολουθεί την ίδια προσέγγιση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή τα private equity, τα ιδιωτικά κεφάλαια δεν μπορούμε να τα συγχαίουμε με τα hedge funds, τα, τα κεφάλαια αντιστάθμισης ε, κινδύνου. Ε, γιατί δεν είχαν καλυφθεί προς το παρόν όταν μιλούσαμε για συστημικούς ε, κινδύνους. Ήταν κάτι διακριτό. Και άρα οφείλουμε να κάνουμε τη διαφοροποίηση ανάμεσα στα διάφορα κεφάλαια που υπάρχουν. Να τονίσω και κάποια άλλα ζητήματα που αναφέρθηκαν ήδη σήμερα. Πρώτον, τα μικρά κεφάλαια. Ή θα πρέπει να έχουμε κατόφλια και να πω επ' αυτού ότι κατέγραψε αυτό που είπε ο εισηγητής ότι δεν είναι υπέρ αυτής της στάσης ούτως ώστε να έχουμε πραγματική και όχι θεωρητική αναλογικότητα. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Ή κατόφλια λοιπόν χρειαζόμαστε ή πραγματική αναλογικότητα. Και είναι περίπλοκο το θέμα, συνιστά πρόκληση. Και γιατί είναι σημαντικό. Διότι εάν δεν κατοχυρώσουμε ευκαιρίε για νεο, ε, ε, νεοεισερχόμενα μικρά κεφάλαια, θα δημιουργήσουμε εξάρτηση από όλο ένα και μεγαλύτερα κεφάλαια. Αντί να κατανέμεται το σύστημα σε διάφορα μικρά ταμεία. Τα μικρά ταμεία όμως είναι πάρα πολύ σημαντικά για τις μικρές επιχειρήσεις, για τις δικές τους επενδύσεις. Οπότε ξαναλέω ή αυστηρή αναλογικότητα που είναι κάτι πολύ δύσκολο ή κατόφλια. Αυτές είναι οι λύσεις. Δεύτερον, ε, οι ε, εταιρείε holding στον τομέα της βιομηχανίας. Πρέπει να είναι σαφέστατοι οι κανόνες, διότι αλλιώς θα ήταν παράδεξο αν ένα τράστ, ένα καταπίστευμα ή ένα holding ε, συμπεριληφθούν τελικά στους κανόνες, γιατί θα αλλάξουμε την ίδια τη φύση αυτών των ομίλων είναι τον όνου κάνευ, κατά τη γνώμη μου, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με αυτό το νομοθέτημα. Τρίτον, οι τρίτε χώρες. Τονίστηκε το θέμα ήδη και δεν θα επιμείνω πολύ. Αλλά ε, επισημαίνω ότι είναι αναγκαίο να το ρυθμίσουμε το ζήτημα για να έχουν ε, εύρυθμες χρηματοπιστωτικές αγορές ε, οι ευρωπαϊκές χώρες για να έχουμε καλά συνταξιδοτικά συστήματα αλλά και για να έχουμε αλλοδαπές επενδύσεις στην Ευρώπη. Δεν είμαι σίγουρος ότι έχουμε ε, επιτύχει το στόχο μας σε αυτό το τομέα. Ε, θα σταματήσω εδώ γιατί δεν έχω και άλλο χρόνο, Πρόεδρε. Νομίζω εξήγησα τα τρία λεπτά. Ευχαριστούμε ο κύριος Μπέλς. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ε, τονίσω ότι ο Ζαμπόλ έκανε εξαιρετική δουλειά και αν λάβουμε υπόψη και την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα ελαττώματα που είχε, τα λάθη που είχε, το οποίο παραδέχεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι δύσκολο να δουλέψουμε με μια γενική προσέγγιση η οποία θα συνοψίζει, αν θέλετε, ε, θα πρέπει να αποτρέψουμε τις αρνητικές συνέπειες για να μην υποσκάψουμε το μέλλον των επιχειρήσεων και να μην καταλήξουμε σε μια υπερβολική συγκέντρωση των, ε, της αγοράς. Το σημείο εκκίνησης ε, της εργασίας ε, για το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έκανε συγκεκριμένε προτάσεις για τα διάφορα επενδυτικά ταμεία. Και το θέμα λοιπόν τίθεται για τις επενδύσεις υψηλού κινδύνου. Και καταλαβαίνω τον εισηγητή που είναι εξαιρετικά διστακτικός. 20 μετοχικά σχέδια που δεν θέλουν να αφήσουν χωρίς ρύθμιση κανένα α, τομέα Και έτσι επαναρχόμαστε στην παλιά συζήτηση για τον συστημικό κίνδυνο και την αρχή της αναλογικότητας. Η καλύτερη λύση ήταν τα εθνικά επενδυτικά ταμεία. Και θεωρώ ότι καλύπτονται οι κίνδυνοι σε ό,τι αφορά τους ομίλους. Άλλες τροπολογίες έχουν γίνει για, για το one size fits all και την ε, προσέγγιση αυτή. Αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να το αποφύγουμε. Η συνοχή με άλλες οδηγία θα πρέπει να εξεταστεί επαρκώς και ο Ζαν Πολ ε, έκανε πολύ καλές προτάσεις στο σημείο αυτό σε ό,τι αφορά το short selling, τις ακάλυπτες πωλήσει, θα ήθελα να υπάρχει μια κατάλληλη λύση η οποία θα καλύπτει όλους τους τομείς. Στο θέμα της μόχλευσης είμαι υπέρ μιας ισορροπημένης ε, προσέγγισης προκειμένου να ε, υπάρχει καλύτερη αντιμετώπιση του κινδύνου που ενέχουν τα hedge funds. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι όπως η καταχώρηση, η εποπτεία, είναι ενδεδειγμένες. Δεν θα πρέπει να θέλουμε να έχουμε ως στόχο την απομόνωση της αγοράς. Και κλείνω με αυτό, αλλά επειδή δεν έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας, θα ολοκληρώσω το σημείο αυτό. Thank you very much. We will have another... Σας ευχαριστώ και θα έχουμε και άλλη ε, ευκαιρία να το συζητήσουμε το θέμα αυτό. Η Άστα Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν χρειάζεται να συγχαρώ τον κύριο Γκοζέ. Θα αρχίσω κατευθείαν τα σχόλια Ξέρετε, χρειαζόμαστε ισότιμη μεταχείριση για τα εναλλακτικά κεφάλαια, είτε βρίσκονται εντό είτε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι η βασική και απλή αρχή. Μπορεί να σα φαίνεται προφανέ αυτό, αλλά στην ουσία περιπλέκονται περισσότερο τα πράγματα σε σχέση με το πεδίο εφαρμογή ε, τη οδηγία. Όλα τα εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια πρέπει να ενταχθούν στην ίδια σειρά κανόνων. Μην ξεχάσετε ότι η οσεκά, τα κεφάλαια μη οσεκά, εξορισμού θα γίνουν εναλλακτικά. Σε αυτήν την λογική θα πρέπει να καλύψουμε με αυτή την οδηγία και τα κεφάλαια που δραστηριοποιούνται εκτός εθνικών αγορών. Εμένα δεν μου αρέσει να βλέπουμε τα πράγματα από εθνική σκοπιά γιατί αυτή η στάση αντιτίθεται στην οικοδόμηση της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών. Θα ήθελα όλα, όλα τα κεφάλαια να υπάγονται στους ίδιους κανόνες. Δεν μπορεί από τη μία να λέμε ότι τα εναλλακτικά κεφάλαια πρέπει να ρυθμιστούν λόγω των συστημικών κινδύνων που επισύρουν και από την άλλη πλευρά να αποκλείσουμε από το πεδίο εφαρμογής όλα τα εναλλακτικά κεφάλαια που ε, είναι αμυγός εθνικά. Ελπίζω να πείσω το Ζαμπόλ για αυτό το θέμα. Ε, για τα εναλλακτικά κεφάλαια τρίτων χωρών ε, το ίδιο πρόβλημα είναι αλλά τίθεται με διαφορετικούς όρου. Προτείνει ο εισηγητή νέο καθεστώς, καθεστώς εθνικών επενδύσεων συν ισοδυναμία. Ωραία. Βάσει αυτή τη πρόταση, τα κεφάλαια τρίτων χωρών μπορούν να κατανεμηθούν ισότιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με καθεστώτα ιδιωτικών εθνικών επενδύσεων, χωρί να χρειάζεται να υπάγονται στου ελαχίστου όρου τη οδηγία, ε, χάρη σε αυτό το σύστημα ισοδυναμία. Αυτό το προσωρινό καθεστώ, συγγνώμη, αλλά είναι προβληματικό. Ελοχεύει μεγάλο κίνδυνο τρέβλωση, ανταγωνισμού, ακόμη και στην αγορά ενό ε, κράτου, ε, γιατί για με, κάποια χρόνια θα υπάρχουν δύο ειδών κεφάλαια ε, θα έχουμε τα κεφάλαια με το διαβατήριο που θα πρέπει να υπάγονται στην οδηγία και από την άλλη θα έχουμε τα κεφάλαια των τρίτων χωρών που δεν θα χρειάζεται να ε, εφαρμόζουν την οδηγία και θα έχουν ως εκ τούτου ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Και ως εκ τούτου αυτό είναι σοβαρό κίνητρο για τα κεφάλαια και τους διαχειριστές να πάνε να εγκατασταθούν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διαβατήριο δεν το αντισταθμίζει αυτό το μειονέκτημα και γι' αυτό, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να οδεύσουμε απευθεία προς μια συμβαστική λύση ναι θέση σε εμπορία των προϊόντων των κεφαλαίων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα υπάγονται σε αυστηρά και ελάχιστα πρότυπα που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως και για τα επενδυτικά κεφάλαια, θέλουμε επίσης η οδηγία να αναγνωρίσει τα αυτοδιαχειριζόμενα κεφάλαια που δεν προσφεύγουν σε διαχειριστική εταιρεία. Όχι να προβλεφθεί εξαίρεση το αντίθετο. Αυτού του είδους οι δομές πρέπει να αναγνωριστούν και να υπαχθούν στην οδηγία. Τέλος, ο ρόλος των θεματοφυλάκων. Πρέπει να αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα στις ευθύνες των θεματοφυλάκων για να αποφύγουμε τα δυσάρεστα που ζήσαμε πρόσφατα, αλλά ας μην υπερβάλλουμε, είναι μία αποτελεσματικό να επομιστούν οι θεματοφύλακες την ευθύνη για επιχειρήσεις για δραστηριότητες που δεν ελέγχουν. Δεν είναι λογικό ε, τους θεματοφύλακες ε, να τους ρυθμίσουμε γενικά γιατί έχουμε τα παραδοσιακά και μη παραδοσιακά ε, εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια και άρα πρέπει να αναδιατυπώσουμε το κείμενο τόσο ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Ε, και είπε ο Ζαν Πολ ότι δεν θέλει η Ευρώπη να είναι ε, ε, οχυρό αλλά ούτε και ξέφραγο αμπέλι. Ελπίζω να με ακολουθήσει στις προτάσεις που έκανα. Ευχαριστώ. Ο Πίτερ. Η Άστριτ με κάνει να γίνομαι πιο ριζοσπαστικός όταν μιλάω μετά από εκείνη αλλά Ζαν Πολ, τι να πω, εξαιρετική εργασία. Νομίζω ότι άνοιξε ένα δρόμο και έτσι θα είναι πολύ πιο εύκολο για μας να σε ακολουθήσουμε. Κινείσαι προς, την, ε, προς τη σωστή κατεύθυνση, μιλάμε για 1660 τροπολογίες στο τομέα της αναλογικότητας έχει μεγάλη σημασία να φτάσουμε σε κάτι καινοτόμο, διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άνοιξε το δρόμο. Υπάρχει συνένεση στο σώμα, αλλά πρόκειται για ένα μεγάλο βάρος που φέρεις εσύ. Και νομίζω ότι η μελλοντική νομοθεσία αρχίζει από εδώ. Μιλήσαμε για πολλές εξαιρέσεις που ε, συρρυκνώνουν την εμβέλεια της οδηγίας. Αυτό που έχει σημασία είναι να εφαρμόσουμε μια νομοθεσία που να είναι αναλογική πραγματικά. Ο Γκούναρ μίλησε για κατόφλια, αλλά νομίζω ότι αν κινηθούμε με κατόφλια θα χάσουμε τη μάχη με το Συμβούλιο, διότι θα πρέπει να ζητήσουμε, να απαιτήσουμε από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εφαρμόσουν ε, έξυπνες λύσεις. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο Ρόμπερτ Γκέμπλξ Goebbels σε σχέση με τις ακάλυπτες πωλήσει οψιών νομίζω ότι θα πρέπει να διέπονται από ένα ιδιαίτερο καθεστώς αν και οι ακάλυπτες πωλήσει δεν είναι κάτι το διαβολικό καθεαυτό. Δεν πρέπει δηλαδή να απαγορευτούν επειδή είναι ακάλυπτες. Έχω υποβάλει τις δικές μου τροπολογίες. Θα ήθελα να προτείνω και τις τροπολογίες της Κάθριν Στάιλερ στο θέμα των τρίτων χωρών, κατανόπροστα που κινείσαι και εσύ ο Ρόμπερτ είπε ότι δεν θέλουμε να είμαστε μια Ευρώπη οχυρό, θέλουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις, αλλά δεν μπορούμε να μην ρυθμίσουμε την αγορά. Γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε μια εξισορρόπηση και γι' αυτό θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα συμβασμό. Το θέμα της αμόχλευσης θα πρέπει να εξεταστεί εκ του σύνεγγης θα πρέπει να έχουμε μία ε, αγορά εποπτείας, έναν πραγματικό επόπτη της αγοράς. Ο Μέιντοφ ε, ε, προώθησε την έννοια των hoodwinking consumers και θα πρέπει εμείς να προστατεύσουμε τους καταναλωτές. Γι' αυτό ε, ε, τόνισα ότι το θέμα των θέματοφυλάκων θα πρέπει να είναι ξεχωριστό από το θέμα διαχείρισης κεφαλαίων. Ε, σε συγχαίρω για την εργασία σου και φαντάζομαι ότι θα φτάσουμε σε έναν απότερο συμβιβασμό. Βίκυ, Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε, Ζαν Πολ, για τα εξαιρετικά σχόλια δεν θα πρέπει να είμαστε οχυρό ή φυλακή και θα πρέπει να το σκεφτόμαστε αυτό όταν ε, μιλάμε και για νομοθεσία σε άλλους τομείς, γιατί μιλάμε για μια παγκόσμια αγορά. Συμφωνώ για την εμβέλεια του εγγράφου, συμφωνώ με τα σχόλια του κυρίου Κλίνς, ότι θα ήταν σκόπιμο να μην ξεχνάμε ότι τα κεφάλαια είναι διαφορετικά τα στοιχεία ενεργητικού είναι διαφορετικά και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε μία ξεχωριστή οδηγία για τα κεφάλαια αντιστάθμισης επιχειρηματικού κινδύνου, δηλαδή άλλο τα hedge funds και άλλο τα ιδιωτικά κεφάλαια. Θα πρέπει να έχουμε μία ξεχωριστή οδηγία για αυτά. Εάν χρειάζεσαι περισσότερο καιρό, θα πρέπει να σου τον δώσουμε. Θα πρέπει να προωθήσουμε αυτή την νομοθεσία ζωτικής σημασίας. Ως προς το θέμα της αναλογικότητας, συμφωνώ μαζί σου θα πρέπει τα ιστορικά κεφάλαια σε ιδιαίτερα αποθεμα... Ε, ταμεία αποθεματικού ή ταμεία παρακαταθήκων θα πρέπει να τα υποστηρίξουμε. Υπάρχει διαφορά μεταξύ μόχλευσης και κίνδυνου. Υψηλή μόχλευση δεν σημαίνει υψηλός κίνδυνος. Κάτι, ένα στοιχείο χαμηλής μόχλευσης μπορεί να ενέχει υψηλό κίνδυνο. Όταν λοιπόν μιλάμε για στόχο αυτής της οδικίας, δηλαδή να σταματήσουμε τον ε, συστημικό κίνδυνο, θα πρέπει να είμαστε σαφείς ως προς αυτό, ως προς τον συστημικό κίνδυνο. Δηλαδή η υψηλή μόχλευση δεν σημαίνει και υψηλός ε, υψηλό κίνδυνο. Όσον αφορά τις ακάλυπτες πωλήσει και τις ακάλυπτες πωλήσει οψιών, στις οψιών υπάρχει διαφορά γιατί μιλάμε για hedge funds, για κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου ως προς τις ακάλυπτες πωλήσει. Νομίζω ότι οι ακάλυπτες πωλήσει θα πρέπει να καλυφθούν από την, από την οδηγία που διέπει τις αγορές. Άρα ίσως για να απλουστεύσουμε τις συζητήσεις θα πρέπει να μιλήσουμε για τις καταχρήσεις, θα πρέπει δηλαδή το θέμα των ακαλύπτων να ε, διέπεται από μια ξεχωριστή ε, ε, οδηγία. Το 1669 ξέρουμε ότι η Έτνα εξεράγει. Όταν μιλάμε λοιπόν για 1669 οδηγίες δεν είναι τόσο δυσίωνες λόγω αριθμού. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να πληγεί η αγορά σε σχέση με τις αγορές, το συνταξιοδοτικό, τη στιγμή που δεν μπορούμε να το στηρίξουμε. Γι' αυτό θα πρέπει να τη ρήτρα 1634, δηλαδή να προσπαθήσουμε να μην έχουμε δυσίων συνέπειες, διότι οι 1669 ε, τροπολογίες ίσως είναι ιδιαίτερα πολλές και να μην μπορούμε να τις διαχειριστούμε ούντο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εμείς από την ομάδα μας ε, θέλουμε να κάνουμε τρία σχόλια ουσιαστικά. Τρία σχόλια. Ε, να συγχαρούμε ασφαλώς τον Ζανπόλ... Ε, για το βαρύ έργο το οποίο έχει επιφορτιστεί σε ό,τι αφορά τις 1669 τροπολογίες όπου ο συνάδελφος ε, κύριος Γκέπελς, ο Σκιώδης, ε, ε, υπέδειξε ότι είναι χρήσιμο να πούμε ότι υπάρχουν και επαναλήψεις, να πούμε ότι υπάρχουν και προγράμματα στους υπολογιστών. Δηλαδή προγράμματα τα οποία μπορούν να συγκεράσουν αν θέλετε κάποια κείμενα τα οποία θα διευκολύνουν το έργο του Ζαν Πολ. Αν μπορούν να γίνουν δηλαδή κάποιες ομαδοποιήσεις των ανθρωπολογιών. Το δεύτερο σημείο το οποίο θα θέλαμε να τονίσουμε ως ομάδα είναι ότι όταν κλείνουν τα φώτα τη νύχτα εδώ στην αίθουσα και ο Ζαν Πολ κλείνει στο δωμάτιο του, να του φέρουμε ένα καφέ για να αντέξει, το οποίο και ελπίζουμε. Και κατά τρίτον, όπως είπε και ο κύριος Γκέμπελς, θέλω να πω ότι ναι, επί της ουσίας ναι, Θέλουμε μια ευφύη ρύθμιση, όπως ακούσαμε, smart regulation, αλλά δεν θέλουμε μια υπερβολικά απλουστευμένη ρύθμιση, η οποία ουσιαστικά δεν θα ρυθμίζει επαρκώς. Γι' αυτό λοιπόν και είπα ότι θα πρέπει να συζητήσουμε το πεδίο εφαρμογή και θα πρέπει να συζητήσουμε και τις επενδύσεις σε τις αλλοδαπές, γιατί ακριβώς ε, συμπεριλάβαμε το θέμα της κυρίας Λούλινγκ. Δεν θέλουμε να υπάρχει αυτή η διαφορά μεταξύ αλλοδαπών και εγχώριων επενδύσεων ούτε να ξεκινήσουμε συζητήσεις για το κατά πόσο υπάρχει λόγος να υπάρχει και να συμμετέχει κανείς στην ευρωπαϊκή αγορά. Κάναμε συγκεκριμένες ε, προτάσεις για όλα τα θέματα, για το short selling, για τα private equities, για το asset stripping. Αυτή θα είναι η, οι βασικοί πυλώνες της ρύθμισης αυτής. Εκεί θα κρυθεί η ποιότητα της ρύθμισης. Αν θέλουμε να αποβάλουμε τα τοξικά στοιχεία, δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να παραμείνουν άλλοτε αυτά τα θέματα. Και υπάρχει και ένα σημείο το οποίο θα θέλα πραγματικά να το τονίσω. Και συνάδελφοι, ναι, να μάθουμε και να πληροφορηθούμε από τα ιδιωτικά λόμπι, εντάξει, αλλά καταφατικά να γνέφουμε δεν επιτρέπουμε. Χτες κάθισα και μία ώρα πάλι άκουγα αυτά που υπόθηκαν για τα δημόσια χρέη. Ε, πρέπει να κοιτάξουμε ποιοι είναι οι παράγοντες, ποιοι είναι οι φορείς οι οποίοι κερδοσκοπούν εις βάρος του δημόσιου χρέους και δεν μπορούμε να γνέφουμε απλά καταφατικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Όπως είπε και ο Ζων Πολ, χρειαζόμαστε ποιοτική ρύθμιση. Thank Σας ευχαριστώ. Ο επόμενος λέει Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά τα διάφορα ταμεία και τις διάφορες επενδύσεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ρυθμίσουμε τόσα πολλά θέματα. Ε, ε, είναι σημαντικό να βρούμε τη σωστή λύση διαπιστώνουμε ότι αυτή η ευρεία και περίπλοκη συζήτηση που κάνουμε για να μπορέσει να οδηγήσει σε ένα καλό συμπερασμό πρέπει να βρούμε μία ισορροπία, γιατί έχουμε πολυάριθμες τροπολογίες. Πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε τρία βασικά σημεία επί της αρχής. Πρώτον, ε, λέξη κλειδί, διαφάνεια. Ενίσχυση της εποπτείας ε, των κεφαλαίων ε, για να μειώσουμε τον κίνδυνο. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, να επομίζονται οι διαχειριστές τις ευθύνες τους και είναι απαραίτητο να μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά ε, οι εποπτικές αρχές για να αντιμετωπίζουν τους συστημικούς κινδύνους. Τώρα, η δεύτερη βασική αρχή είναι η αναλογικότητα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, δηλαδή οι διάφορες ρυθμίσει θα πρέπει να προσαρμοστούν στου πραγματικού κινδύνους για τα διάφορα κεφάλαια που υπάρχουν, γιατί αυτοί οι κίνδυνοι επηρεάζουν ολόκληρη την κοινωνία. Πρέπει να ρυθμίσουμε, λένε και αυστηρότερο όσο αυξάνονται και οι κίνδυνοι. Τα μικρά κεφάλαια επισύρουν μικρότερους κινδύνους σε σχέση με τα μεγαλύτερα. Και ε, ε, μπορεί κανείς να προτάξει σωστά επιχειρήματα σχετικά με τα κεφάλαια private equity. Ε, αν πει ότι έχουν αυστηρότερο σύστημα σε σχέση με τα κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου. Τρίτον, ο προστατευτισμός στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε διάφορες ε, τροπολογίες υπάρχουν ανησυχητικά στοιχεία ε, θα πρέπει να ρυθμίσουμε την δραστηριότητα των διαχειριστών ε, στην Ευρώπη, χωρίς όμως να κλείσουμε και την πόρτα σε τρίτες χώρες. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε ισορροπία στις διάφορες ε, ρυθμιστικές αρχές και για να τα καταφέρουμε θα πρέπει να έχουμε κατοχυρώσει ε, κρατές αρχές στις οποίες θα βασιστούμε για τις μελλοντικές ρυθμίσεις. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστούμε. Ε, κυρία Τζόρι είναι εδώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ θα ήθελα να κάνω ορισμένα σχόλια. Όπως είπε και ο προλαλής σας και όπως είπε και ο Γκούναρ θα πρέπει να έχουμε τα 100 εκατομμύρια κατόφλι διότι αν δεν υπάρχει αυτό το κατόφλι τότε οι διαχειριστές κεφαλαίων μεσαίου μεγέθους θα πρέπει να κινηθούν σε τρίτες χώρες για να αποφύγουν το γραφειοκρατικό φόρτο αλλά νομίζω ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει μια τέτοια παθητική στάση, διότι θα πλήξει τους εθνικούς ε, προϋπολογισμούς και τους εθνικούς διαχειριστές. Δεύτερον, ως προς την αρχική πρόταση, η αρχική πρόταση δεν ε, περιλαμβάνει ειδικούς κανόνες για διάφορα είδη κεφαλαίων δεν διαχωρίζει τα είδη κεφαλαίων που θα διέπονται από ρύθμιση ή αρμπιτράζ. Νομίζω λοιπόν ότι θα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ανταγωνιστικής μειονεξίας και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί και δεν υπηρετείται έτσι σε σχέση με τους επενδυτές λιανικής, ακόμα και στις δευτερεύουσες αγορές, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να μπορούν να έχουν μερίδιο σε εναλλακτικά κεφάλαια, διότι κατά αυτό το τρόπο θα μπορέσουν να υπεκφύγουν των κανόνων αυτών. Τέλος, στις τροπολογίες μου ε, πρότεινα έναν δίκτυ επιπρόσθετου ή συνολικού κινδύνου, όπου η υψηλή μόχλευση, ιδιαίτερα ως προς τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και αντιστάθμισης, θα μπορέσουν να συσσωρευτούν, δηλαδή να ζούμε συνολικά υπομορφή δίκτυ. Η Επιτροπή είναι σε θέση να αποφασίσει για το δίκτυο αυτό και οι υποπτικές αρχές θα πρέπει να επέμβουν τη στιγμή που τα κεφάλαια έχουν υπερβεί αυτό τον δίκτυο και έτσι θα μπορούν να τύχουν διαχείρισης σε καθημερινή βάση ως προς τους εμπλεκόμενους κινδύνους. κυρία Αντρέσεν, ζητήσατε τηλεφωνικά το λόγο σε αυτή τη συζήτηση. Θέλετε να λάβετε κι εσείς το λόγο στα AIFM για τρία λεπτά maximum. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γκοζές για την εργασία του. Η πρόταση αυτή ανέκυψε μετά από την κρίση του 2009 πριν βεβαίως υπήρχε μεγάλη ανησυχία για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τα hedge funds είναι υπόλογα για την κατάρρευση του τρόπου διαχείρισης κεφαλαίων και μετά είχαμε τα γεγονότα του 2008 και 2009 και θεωρούσαμε ότι έπρεπε να περιορίσουμε τη μόχλευση. Θυμόσαστε τη μεγάλη μόχλευση του LTCM. Θα πρέπει να ορίσουμε το γεγονός ότι η μόχλευση των hedge funds έχει μειωθεί εάν λάβουμε υπόψη το LTCM. Και νομίζω ότι σήμερα έχουμε να κάνουμε με μία ε, κίνηση η οποία ήρθε πολύ αργά. Τη στιγμή που έπρεπε να έχουμε όρια ε, μόχλευσης θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη την κατάσταση των τραπεζών που μας οδήγησε για το που είμαστε σήμερα. Θα ήθελα να σας πω ότι κανένα hedge fund δεν ζήτησε διάσωση και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι κατέρευσαν οι παγκόσμιες οικονομίες. Και το δεύτερο σημείο είναι ότι αυτή η οδηγία που θέλει να διέπει τα πάντα δεν καλύπτει μόνο τα στοιχεία ενεργητικού. Καλύπτει τα, ε, τα ταμεία καταπίστευσης και τα κεφάλαια, καθώς και τα hedge funds. Υπάρχουν όμως πολλά είδη κεφαλαίου εδώ. Εγώ έχω υποβάλει μία τροπολογία για να μην λαμβάνω υπόψη το καταπίστευμα, τα καταπιστεύματα, τα οποία είναι διαφορετικά από τα hedge funds που πλήττονται από αυτή τη ρύθμιση. Επίσης έχουμε έχω υποβάλει μία τροπολογία για να διπλασιάσουμε το κατόφλι, αν και βλέπω ότι άλλοι ε, προέτρεξαν ως προς αυτό και τις υποστηρίζω. Ως προς τα κεφάλαια τρίτων χωρών, οι νέες προτάσεις της Ισπανικής Προεδρίας οδηγούν σε μία προστατευτική ρύθμιση της αγοράς, αφήνοντας την αγορά σε κεφάλαια εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι ο προστατευτισμός αυτός θα μας πλήξει. Ως προς την πληθώρα τροπολογιών, τη σωρία τροπολογιών, η πρόταση Επιτροπής δεν είναι ικανοποιητική. Διαφορετικά δεν θα είχαν ανακύψει τόσες πολλές τροπολογίες, σχεδόν 1.700. Θα ήθελα να αποστείλουμε την πρόταση στην Επιτροπή και να ζητήσουμε αναδιατύπωση, λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Εγώ είμαι η τελική ομινήτρια. Θα ήθελα να πω ε, δύο-τρία λόγια, γιατί κάποια από τα θέματα που ήθελα να αναφέρω έχουν καλυφθεί, αλλά κάποιοι τομεί στην οδηγία αυτή αποτελούν, αν θέλετε, σημεία που επικαλύπτονται με υφιστάμενες ε, οδηγίες σε ό,τι αφορά τις ακαλύπτες ε, πωλήσει, το naked short selling και τα παράγωγα και στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να καλυφθούν από την κατάχρηση των αγορών μπορεί να διαμορφώσουμε καλύτερη εντύπωση για τις κερδοσκοπικές δραστηριότητες όταν θα υπάρξουν τα αποθεματικά για την ε, ναι, την εκαθάριση παραγωγών. Θα με ανησυχεί ιδιαίτερα επίσης το ότι δεν επικρατούν ίσως ε, ίσοι όροι για διάφορα είδη ιδιωτικών επιχειρήσεων. Αν, ε, για παράδειγμα, ανήκει κανείς σε private equity, δεν είμαι σίγουρος, σίγουρη ότι υπόκειται κανείς στους σωστούς κανόνες. Θα ήθελα λοιπόν να κοιτάξουμε και το εταιρικό δίκαιο και να βρούμε μέτρα τα οποία θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε. Όσο συνειδητοποιούμε νομίζω πού υπάρχουν αυτές οι επικαλύψεις και όπως, ε, όσο προσεγγίζουμε αυτές τις επικαλύψεις με ευθύ τρόπο, νομίζω ότι θα αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά και ελπίζω να καταφέρουμε να συνεργαστούμε επικοδομητικά με τον εισηγητή. Δεν θα μακρηγορήσω, θα δώσω το λόγο στον Ζαν Πολ για να συνοψίσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τα καλά τους λόγια και για τη συμπόνια που δείχνουν ε, για όσα πρέπει ακόμη να κάνω. Σίγουρα με την ε, αγαστή κατά πως φαίνεται συνεργασία ε, που θα έχουμε στο μέλλον θα καταφέρουμε να βρούμε φυείς λύσεις. Θα ήθελα να απαντήσω σε ένα ή μία συνάδελφο, μία συνάδελφο στην Άστριντ που με εγωιτεύει ε, όπως πάντα. Ε, μάλλον δεν έχεις διαβάσει άστρε τις τελευταίες μου προτάσεις, γιατί δεν απέχουν και τόσο πολλοί απόψεις μας. Ε, οπότε, αν θέλεις, ε, μπορούμε να τα πούμε κατηδίαν για να συγκλίνουν οι απόψεις μας. Λοιπόν, ευχαριστώ τους συνάδελφους. Ευχαριστώ για τη βοήθειά σας, είμαι στη διάθεσή σας και ζητήστε μου ραντεβού, θα συναντηθούμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ευχαριστώ. Διαδικαστικό. Πρόεδρε, φαντάζομαι ότι θα περάσουμε τώρα στις ψηφοφορίες. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω, επειδή έχουμε τόσα πολλά θέματα και επειδή ε, δεν έχουμε ακόμα διοργανωθεί στην ομάδα μας, να κάνουμε μία, ένα μικρό διάλειμμα, τρία ως πέντε λεπτά, για να μπορέσουμε μετά να προχωρήσουμε χωρίς καθυστέρηση στην ψηφοφορία. Συμφωνείτε. Ναι, συμφωνώ λέει η Πρόεδρος. Ε, καλή ιδέα. Πέντε λεπτά διάλειμμα. Θα ήθελα απλά να τονίσω ότι η δεύτερη συζήτηση θα, για το θέμα του, I, του AIFM των διαχειριστών οργανισμών Ανατολικών επενδύσεων μπορεί να γίνει το απόγευμα της 17ης Μαρτίου. Πέντε λεπτά διάλειμμα όμως. Νομίζω ότι πέρασαν τα πέντε λεπτά, λέει η πρόεδρο. Ελπίζω να καταφέρετε να ανασυντάξετε τι δυνάμεις σα, Παρακαλώ καθίστε. Φαίνεται ότι λείπει ακόμα κόσμος. Παρακαλώ, καθίστε. Θα ξεκινήσουν οι ψηφοφορίες, λέει η Πρόεδρο. Ζητήσαμε να φέρετε μαζί τις ε, κάρτες ψηφοφορίας. Ελπίζω να τις έχετε λοιπόν όλοι μαζί. Να υπενθυμίσω ότι είναι μάλλον δύσκολο να ολοκληρωθούν ε, γρήγορα οι ψηφοφορίες. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τις κάρτες μας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τις ψηφοφορίες. Καθίστε παρακαλώ. Πρώτη έκθεση. Η έκθεση για την έκθεση για την ετήσια δήλωση για την Ευρωζώνη το 2009 και τα δημόσια οικονομικά. Τροπολογία 1. Για την αιτιολογική σκέψη Α. Παρακαλώ υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. Τροπολογία 2. διλογικη σκέψη αλφα-αλφα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο του της σκέψης Β. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. αρχικό κείμενο για τη λογική σκέψη D υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ή. E, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. F. Αρχικού κειμένου υπέρ. Κατά. Αποχές Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά βλέπω ότι κουράζονται τα χέρια. Να περάσουμε στην τελική σκέψη G. Συμβαστική α, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να περάσουμε στην τροπολογία 5, λοιπόν. Τροπολογία 5, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία. Ε, τελική σκέψη α Αι συγγνώμη, συμβαστική B, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 7, υπέρ. Ναι, ναι, ναι, αποφασίσατε, υπέρ. Κατά, άποχες, εγκρίνεται. Συμβαστική C, υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται. Και στην περίπτωση λοιπόν αυτή έχουμε την τροπολογία υπαριθμών 8. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεν είμαι βέβαιη. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψήφισατε όλοι. Ψήφισατε όλοι παρακαλώ. Νομίζω ότι ο αριθμός θα πρέπει να είναι προς τα κάτω. Δεν ξέρω, δοκιμάστε αν θέλετε το επόμενο μηχάνημα. Ωραία, λοιπόν, τώρα ψηφίσαμε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Ο Σάντσος έχει πρόβλημα. Εγκρίνεται. 25 υπέρ 18 κατά. Um, amendments 9, 10 fall. So now we go to amendment 11. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Θα πρέπει να το ελέγξουμε και αυτό. Για την τροπολογία 12, ηλεκτρονική ψηφοφορία, παρακαλώ, έναρξη ψηφοφορία. Oh, do wish my group would signal what I'm supposed to be doing, please. Votes closed. Πέρας. That's adopted. Uh, amendment Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική D. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 και 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ή e. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε λοιπόν στη συμβαστική F. Σε τμήματα ψηφοφορία στο πρώτο τμήμα ένα κείμενο που δεν περιλαμβάνει τις λέξεις ε, που βλέπετε μπροστά σας από considers μέχρι food prices. Η πρώτη ψηφοφορία λοιπόν είναι για το σύνολο του κειμένου χωρίς αυτό το κομμάτι. Παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Στο δεύτερο τμήμα είναι οι λέξει που σα διάβασα. Υπέρ, παρακαλώ, του τμήματο αυτού. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας κάνουμε έναν ηλεκτρονικό έλεγχο. Έναρξη ψηφοφορίας. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Και περνάμε στη συμβαστική G, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στην 42, τροπολογία 42, υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές, πολύ φοβάμαι. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 42, παρακαλώ, τροπολογία 42. Right. The vote is closed. Πέρας That's rejected. Απορρίπτεται. Έχατε κάποιο πρόβλημα με την ε, κάρτα σας? Έχουμε λοιπόν τρεις επιπλέον ψήφους. Έχουμε σωστό αριθμό ψηφισάντων, λέει πρόεδρο. Σαν Πολ. Ε, μία ερώτηση. Μπορούμε να ελέγξουμε πόσοι ψηφίζουν. Παρακαλώ. Ε, να δούμε αν εκπροσωπούνται σωστά τα πολιτικά κόμματα. Ε, η κυρία Λούλινγκ, ο κύριος Κάρας. Κύριε Μακάλο, έχετε την κάρτα σας. Ναι, δεν λειτουργεί. Για δοκιμάστε σε κάποιο άλλο μηχανάκι, σε μια άλλη συσκευή. Δεν λειτουργεί. Κύριε Κάρας, η δική σας η κάρτα δουλεύει. Έχει ολοκληρωθεί η ψηφοφορία. Ωραία, να ξανανοίξουμε παρακαλώ την ψηφοφορία για το θέμα αυτό. Για την τροπολογία 42, παρακαλώ, ξανά ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Στην ίδια ψηφοφορία, επαναλαμβάνουμε την ίδια ψηφοφορία. Έναρξη ψηφοφορίας για την 42, παρακαλώ. Έχουμε δύο προστίκες. Ψηφίζει και η κυρία πίσω σας βλέπω. Κυρία Λουλίνγκ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Χάρη στην κυρία Λούλινγκ. Εγκρίνεται, ναι, εγκρίνεται. Τροπολογία 43 και 44. Φαίνεται, φαίνεται αν ψηφίζουν υπερβολικά πολλά άτομα. 45 παρακαλώ. 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 46. Υπέρ. κατά άποχες έλεγχος παρακαλώ ηλεκτρονικός έλεγχος για την 46 Um, could I ask the Να ζητήσω από την ομάδα της Άλντε να μας... Oh. μας πει ποιος ψηφίζει. Πρόεδρε, μπορείτε να έρθετε να ψηφίσετε με εμά αν δεν βρίσκετε άλλη θέση. Δυστυχώ. ξέρετε τώρα, από το ΕΛΚ έχουμε ένα παραπάνω από ό,τι πρέπει. Ζαν Πολ, η ομάδα σας, σε κάποιο είναι... Κάποιος ψηφίζει που δεν έπρεπε να ψηφίζει. Ποιο είναι? Εντάξει λοιπόν τώρα. Να ψηφίσουμε. Πείτε μου, πείτε μου, γιατί κανείς δεν μου έδωσε κατάλογο ψηφοφορίας. Πείτε μου λοιπόν. Αν είσαστε υπέρ ή κατά. Ωραία, εντάξει, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Μα πού, πού είμαι. Ό,τι θέλω κάνω, λέει η πρόεδρος. You had one too many on the η κάρτα σας ε, περίσσευε μία κάρτα. Ψήφιζε ένας παραπάνω. Ναι, αλλά έχετε αρκετές κάρτες οι οποίες λειτουργούν. Well, Μα σα είχα πει να έρθετε να ψηφίσετε με τις κάρτες σας. Εγκρίνετε, εν πάση περιπτώσει. Δεν, εγώ θα προχωρήσω, δεν έχω κάτι άλλο να κάνω. Ψηφίζουμε τη συμβιβαστική age. Υπέρ παρακαλώ. Συμβιβαστική age. Χωρίς τη λέξη πρώτο τμήμα current account. Υπέρ παρακαλώ. Στο πρώτο τμήμα χωρίς τις λέξεις current accounts. Κατά. Αποχές εγκρίνεται με τις λέξεις current accounts τώρα. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Μα δεν σηκώνετε τα χέρια σας. Άρα θα πρέπει να το ελέγξουμε. Να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα. Έτσι ε, να κάνουμε, δεν θα τη βγάλουμε όλη την ημέρα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Has everybody voted? Right, Ψηφίσατε όλοι. Now people are putting their hands up. That's carried. Εγκρίνεται λοιπόν να περάσουμε στην 52. Τροπολογία 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική I. Σε τμήματα. όλο το κείμενο χωρίς την φράση including the setting up of new mechanism. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με την φράση αυτή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική J λοιπόν τώρα. Υπέρ. Συμβιβαστική J. Υπέρ. Κατά. αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Να ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά για την συμβαστική J. Έχουμε και δυσκολίες με την συσκευή εδώ, στο Προεδρείο. Το ΕΛΚ ψηφίζει σωστά. Όχι, περισσεύει ένας από το ΕΛΚ. Χωρίς την Άστριτ. Ναι, αλλά πρόεδρε, ψηφίσω εγώ στη θέση της κυρίας ε, Λούλινγκ. Ναι, αλλά παρόλα αυτά περισσεύει ένας, ο κύριος Μπούλμαν. Πρόεδρε, το θέμα δεν είναι να ορίσουμε μόνο το θέμα, μάλλον το θέμα του αν ψηφίσει σωστό αριθμό των ομάδων δεν εξαρτάται από την ομάδα, η πρόεδρος το καθαρίζει. Και γι' αυτό θα θέλα αυστηρά να ψηφίζουν μόνο όσοι έχουν δικαίωμα ψήφου. Δεν ε, καθορίζει η ομάδα αν ε, ψηφίζουν αρκετοί ή όχι. Όχι, όχι, λέει η Πρόεδρος. Εγώ το καθορίζω. Εδώ η συσκευή μου λέει πότε ε, λειτουργούν υπερβολικά πολλές κάρτες από μία η ομάδα ή όχι. Κάποιες υπερβολικα πολλε λοιπόν έχω μια τέτοια ένδειξη σφάλματος, κάποιες ενδειξη σφαλματο Εδώ οχι Ε, το ελέγχουμε. Βλέπω λοιπόν ότι περισσεύει μία κάρτα για το ΕΛΚ. Ο κύριος Λάμεν. Ναι, θα ήθελα να δώσω δίκιο στην Πρόεδρο. Δεν είναι δυνατόν να αποφασίζουν η ομάδα ποιος ε, θα ψηφίζει. Η Πρόεδρος θα αποφασίζει και όχι ο συνάδελφος Μπούλμαν. Ωραία, λέει ο Πρόεδρος. Ναι, συγγνώμη. Τώρα, εντάξει. Τώρα είμαστε εντάξει, λέει ο Πρόεδρος. Ε, ψήφιζα ως τώρα, αλλά αν περισσεύω, να σταματήσω να ψηφίζω. Ωραία, λέει η πρόεδρο. Τώρα, εντάξει, στέκει ο αριθμό των πέρα ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Και θα ήταν πολύ πιο απλά τα πράγματα αν σηκώνετε τα χέρια σα. Συμβαστική J, λοιπόν, να περάσουμε στην τροπολογία 60 τώρα. 60, 61, 62. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 63 60, έως 66 καταπίπτουν. Συμβαστική K, κάπα, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική L, υπέρ, κατά. Συμβαστική L, υπέρ, κατά, αποχές Απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε στην τροπολογία 71 και 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Θέλετε έλεγχο, να το ελέγξουμε για την 71 και την 72, παρακαλώ, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Όντως εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβαστική M, μη, υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 79, τροπολογία 79, υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 80 που είναι συμβατή. Παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται θεωρώ. Να το ελέγξω αν θέλετε. Για την τροπολογία το παρακαλώ. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Όντω εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβαστική νη. Εν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και περνάμε στην 88 παρακαλώ τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται αλλά λίγα χέρια σηκώθηκαν. 89 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 91 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 97 παρακαλώ. Με προφορική τροπολογία. Για να συμπεριληφθούν οι λέξει στο άρθρο 136 του. Χρειάζεται κανείς διευκρινήσεις, υπάρχουν ενστάσεις. Άρα λοιπόν το σύνολο της τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Στην 98 παρακαλώ. Τροπολογία 98. Και εδώ έχουμε προφορική τροπολογία. Να αντικατασταθούν οι λέξεις disrespect με το κείμενο που βλέπετε μπροστά. Στον κατάλογο ψηφοφορία, δεν θα το διαβάσω. Υπέρ της προφορικής τροπολογίας κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ο όμικρον. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική π. Και αν φαίνεται ότι υπάρχει μια αλλαγή τελευταία στιγμή. Έχετε μπροστά σα την αλλαγή αυτή. Σε τμήματα λοιπόν ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα Χωρί το κείμενο που βλέπετε από το points out μέχρι the spirit. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με τις λέξεις αυτές, τη διατύπωση αυτή υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίφθηκε η διατύπωση. Α, είναι και το τρίτο τμήμα βέβαια. Για το The Spirit. Στο τρίτο τμήμα, για τη διατύπωση αυτή, παρακαλώ. Υπέρ τη συμπερίληψη τη διατύπωση αυτή. Κατά. Αποχές. Ωραία. Δεν πέρασε και το spirit. Περνάμε στην τροπολογία 107. Υπέρ. 107 παρακαλώ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται από τα χέρια που, ίδια, που είδα. Αν δεν τα σηκώνετε, τι να κάνουμε. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές. Αν το ΕΛΚ θέλει να ψηφίσει, να σηκώνει τα χέρια του παρακαλώ. Γιατί δεν βλέπω τίποτα. Υπέρ για την 109 παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 110 υπέρ. Α, συγγνώμη, έχει καταπέσει. Για την συμβαστική Q αναφέρεται ότι οι σοσιαλιστές θέλουν να γίνει προφορική τροπολογία, να αναφέρεται κάποια κράτη-μέλη, να μην υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά στην Ελλάδα. Ε, καμία ένσταση, υποστήριξη της προφορικής τροπολογίας αυτής. Ο Hans Peter Martin. Είχα ζητήσει το λόγο για το θέμα αυτό και θα ήθελα να πω ότι με προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι προετοιμάζουμε μία τροπολογία η οποία είναι ε, ίδια με τη δική μου τροπολογία εκτός από δύο λέξεις. Και μετά έχουμε συζητήσει ε, καν το θέμα αυτό. Τι δηλαδή, αυτό το κοινοβούλιο λειτουργεί σε δύο επίπεδα. Δεν συμφωνώ καθόλου σε ό,τι αφορά δηλαδή την προετοιμασία των τροπολογιών. Κύριε Μπούλμαν, δυστυχώς δεν μπορώ να εκφραστώ επ' αυτού. Δεν με έχουν ενημερώσει για αυτό που είπε ο συναδελφός Χάνς Πέτερ Μάρτιν, αλλά θα ήθελα να πω ποια είναι η δική μας η θέση για τη συμβιβαστική Q. Γιατί υπάρχει παράδοση εδώ στο Κοινοβούλιο να μιλάμε για προβλήματα, αλλά να μην κατονομάζουμε συγκεκριμένες χώρες, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν περισσότερες χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Αυτή είναι η αιτιολόγηση της πρότασής μας. Δεν θέλουμε να ξεκινήσουμε πολιτική συζήτηση, απλά θα θέλαμε να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχιστεί αυτή θα συνεχιστεί αυτή η παράδοση του Κοινοβουλίου και γι' αυτό λοιπόν έχουμε κάνει αυτή την προφορική τροπολογία στο συμβαστική Q. Σίλβη. Πρόεδρε, δεν νομίζω ότι είναι πολιτικό το θέμα. Είναι ουσιαστικό, έτσι. Τα στατιστικά προβλήματα είναι πολύ σοβαρότερα στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Um, Άρα υποβάλλεται ένσταση στην προφορική τροπολογία. Υποβάλλεται επίσημα ένσταση, Σίλβη. Ναι, γιατί αν υποβάλλεται ένσταση, καταπέπτει, καταπίπτει η προφορική τροπολογία. Σίλβη, παρακαλώ με το μικρόφωνο σας. Ναι, μάλιστα, είναι επίσημη ένσταση. Λοιπόν, το χρειαζόμαστε αυτό για τα πρακτικά. Ωραία, λοιπόν, θα ψηφίσουμε με την ε, συμπερίληψη της Ελλάδας. Υπέρ της συμβαστικής Q, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται η γραμματεία μου υπέδειξε ότι έχω ξεχάσει κάποιες τροπολογίες, η 91. η 92 και 93 επίσης θα πρέπει να ψηφιστούν μετά την 91. 92 λοιπόν, η οποία είναι συμβατή με την 91. Παρακαλώ λοιπόν στη σελίδα 14 του καταλόγου ψηφοφορίας και να ψηφίσουμε την 92 του κυρίου Gong. Παρακαλώ υπέρ. Την 92, την 92 λέει ο πρόεδρος. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Καταπίπτει η 93. Ωραία. Ωραία και επιστρέφουμε λοιπόν στην 112. Υπέρ. Υπέρ. Στην 112 κατά αποχές εγκρίνεται. Η 213 υπέρ κατά εγκρίνεται. 114 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική R υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική S. Σε τμήματα, σε τρία τμήματα συγκεκριμένα. Το πρώτο τμήμα, παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, με τη διατύπωση που βλέπετε, υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα. Με τη διατύπωση που βλέπετε. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Περνάμε στην τροπολογία 126 υπέρ. Κατά. Παρακαλώ ηλεκτρονικός έλεγχος για την 126. Πέρας. And that's rejected απορρίπτεται 127 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται 128 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται αρχικό κείμενο στις παραγράφου 29 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται συμβιβαστική ταφ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 130 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 131 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 132 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 130 τρία σε δύο τμήματα παρακαλώ. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Νομίζω ότι ανάποδα πρέπει να το κάνουμε. Στο πρώτο τμήμα είναι ψηφίζουμε αν είμαστε υπέρ της διατύπωσης. Άρα, πρώτο τμήμα, παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Για τη διατύπωση που βλέπετε μπροστά σας. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Και αυτό εγκρίνεται. Ή 134 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 135 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 137 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 138 υπέρ. Κατά. Αποχές. να το ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά για την 138 έναρξη ψηφοφορίας. Votes closed. Πέρας. That falls because it's 23. Καταπίπτει 23 υπέρ και 23 κατά. I'm glad I said I couldn't tell, I was right something. Για την 139 με προφορική τροπολογία για να διαγραφεί η λέξη expeditious, υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. Η 140, υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. 141, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 142 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε παρακαλώ για την 142. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται με μία ψήφο. 143 καταπίπτει. Περνάμε λοιπόν στην 144 υπέρ. Τι έγινε? Σχόλια εκτός μικροφώνου του κυρίου Μπούλμαν. Α, δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. Εντάξει. 144. υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 145 υπέρ. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα θα ψηφίσουμε το κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Παρακαλώ με τις κάρτες. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Α, πάλι από το ΕΛΚ περισσεύει ένας. Πέρας ψηφοφορίας.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 Sorry, the, the vote. Συγγνώμη. Ε, έκθεση της Σοφία Ιντεβέλτ, έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2008, τροπολογία 1 από την Ήτρε. Ποιοι είναι υπέρ, παρακαλώ, κατά αποϊχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 της ΣΥΜΚΟ, υπέρ Ζητώ συγγνώμη, πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία 14. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Ε, ε, χρειάζεται να ψηφίσουμε και για το πρωτότυπο το 14 να ρωτιέται η Πρόεδρος. Μάλιστα. Υπέρ παρακαλώ για το 14. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15 με προφορική τροπολογία του κυρίου Φέρμπερ σε δύο τμήματα. Πρώτα θα ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία. Ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εμπλακεί στη διαμόρφωση των φορολογικών πολιτικών. Έτσι, συμφωνείτε, ναι. Υπέρ παρακαλώ, για την προφορική τροπολογία ψηφίζουμε κατά αποχές εγκρίθηκε. Τώρα έχουμε τμηματική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα συμπεριλαμβανομένη προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχέ. Απερίφθη. Τμήμα 2. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 16. Κατά τμήματα δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα. Ε, ε, ελέγχουμε ποια σειρά, έτσι, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίθηκε. Και το δεύτερο τμήμα τώρα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 17, υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. 18 τώρα με προφορική τροπολογία του Σάντσες Πρεζέντο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα τι πρέπει να ψηφίσουμε. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4, ΉΜΚΟ. υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική Α, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 23, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ Ζητώ συγγνώμη δίκαιο. έχετε παράγραφος 6 πρέπει να το ψηφίσουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3 ε, τη ΣΥΜΚΟ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 4, Ήτρε, με προφορική τροπολογία του εισηγητή. Ε, γίνεται δεκτή η προφορική τροπολογία, έτσι φαίνεται, υπέρ, κατά, αποχές, ε, ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ξέρετε, αν σηκώνετε, ε, τα χέρια σας, ε, θα με διευκολύνατε πάρα πολύ. Τροπολογία 5, ήτρε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2, ΙΜΚΟ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3, της ήτρε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10 Τη Ήτρε. Υπέρ. Κατά. Κατά. Απορρίπτεται. τριακοστή πρώτη υπέρ. Κατά. Αποχές. Ζητώ συγγνώμη, επαλήθευση, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 31η. Ε, Ψηφίστε παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίθηκε. Ναι. Ε, 39. Ε, 29 υπέρ. Όχι, σαφέ είναι. 29, υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχο παρακαλώ. Γιατί έγινε ξεχωριστή ψηφοφορία στην ομάδα. Για την 29 ψηφίστε ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 5 τη ΣΥΜΚΟ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25 τώρα. Κατά τμήματα παρακαλώ. Με προφορική τροπολογία από τους φιλελευθέρους ε, για το δεύτερο τμήμα. Ε, πρώτα ψηφίζουμε για το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ζανπόλ. Δεν είμαι σίγουρη. Εκτός μικροφώνου. Παρακαλώ, ανάψτε το μικρόφωνο σας για να σας ακούμε. Συγγνώμη, ε, στον κατάλογο έχουμε κάνει τόσες πολλές αλλαγές που δεν ξέρουμε τώρα πού έχουμε φτάσει για την 25. Μιλάτε 6α νέο, για αυτή ψηφίζουμε. Με ψηφοφορία κατά τμήματα που ζήτησαν οι φιλελεύθεροι. Θα σας διαβάσω αυτά που έχω στο δικό μου τον κατάλογο. Τμήμα 1 λέει τονίζει ότι αποσιοποιητικά μέχρι το πολιτιστική προστασία. τμήμα 1 λοιπόν τις 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτωται. Τμήμα 2. Εδώ υπάρχει η προφορική τροπολογία που προτείνει. Ε, ε θεωρεί ότι είναι απαραίτητο μπλα μπλα μπλα κτλ. Και, και δημόσια οικονομικά. Αυτό προσθέτουμε. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα λέει, αν η προφορική τροπολογία γίνει δεκτή, έτσι έγινε. Πολύ ωραία, τελειώσαμε. Συμβαστική γάμα υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Τροπολογία 28 σε δύο τμήματα. Το πρώτο takes the view, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, points out και τα λοιπά. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ε, τροπολογία 32, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 33, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 34 ε, καταπίπτει 35 παραμένει υπέρ It says here 34 Μα λέει 34 κατά πίπτη αν εγκριθεί η 32, έτσι δεν είναι. Είναι συμβατή με την 33 αλλά όχι με την 34. Οπότε τώρα έχουμε περάσει την 35 που είναι συμβατή γενικότερα με όλες. Λοιπόν, υπέρ για την 35 κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ο πρωτότυπο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, ηλεκτρονικός έλεγχος αν θέλετε για 39. Ψηφίστε παρακαλώ. Everybody voted. Votes closed. Πέρας. Εγκρίνεται. Uh, amendment 40. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, συμβαστική δέλτα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. μου λένε εδώ ότι ο εισηγητής ε, θέλει να ψηφίσουμε τη 34 ε, για να συμπληρώσουμε τη συμβαστική δέλτα. Όχι, τη 44, συγγνώμη. Ωραία, υπέρ, κατά. Αποχές. Μπορείτε. Τώρα 45 υποθέτω. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 46, 47 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το πρωτότυπο τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 50 υπέρ. Καταπίπτει, καταπίπτει. Και όλες οι υπόλοιπες. Πού φτάνουμε. Στην 54 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το πρωτότυπο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60. Έχει ήδη εγκριθεί. Δεν ψηφίζουμε. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, απορρίπτεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα reiterates μέχρι το tax base υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα likewise μέχρι το competition υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ κατά αποχές ε, ηλεκτρονικός έλεγχος ε, για την 67 παρακαλώ ψηφίστε Πέρας. Amendment 68. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το πρωτότυπο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 70. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 71. Υπέρ. Α, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το πρωτότυπο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 73. Υπέρ. Κατά. Αποχές Two parts, 73. Δύο τμήματα. Δεν το λέει ο δικός μου κατάλογος. Θα μπορούσε κάποιος να μου εξηγήσει τι συμβαίνει. 73 in two parts. Rapporteur. Ο εισηγητής, Jean-Paul. Ας μου εξηγήσει κάποιος ποια είναι τα δύο τμήματα, γιατί στο δικό μου τον κατάλογο δεν ε, αναγράφεται. Πρέπει κάποιος να το προτείνει για να ψηφίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Παρακαλώ, διευκρινίστε το. Ähm, λοιπόν, το πρώτο κομμάτι welcomes μέχρι το underlines και το δεύτερο τμήμα underlines και μετά. Στο underlines θα γίνει η διχοτόμηση, εντάξει. Okay. Yeah. Έχει Ανωτελεία. To, Okay. Right. This, this... Μάλιστα. Λοιπόν, πρώτο τμήμα. Regards positively και τα λοιπά μέχρι τις κατευθυντήριες ε, γραμμές ε, στον τομέα της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέχρι τις SMEs δηλαδή είναι το πρώτο τμήμα και με τα underlines ε, τονίζει ότι η διευκόλυνση της χρηματοδότησης είναι αναγκαία για την προαγωγή του ανταγωνισμού. Μέχρι το competition δηλαδή το δεύτερο τμήμα. Η πρώτη και η δεύτερη πρόταση συνιστούν το πρώτο και το δεύτερο τμήμα αντίστοιχα. Υπέρ. Για το πρώτο τμήμα παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Από το underlines. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα εγκρίθηκε μόνο και τώρα έχω χαθεί εντελώς, λέει η πρόεδρος. Σόφη, διαδικαστικό χτες ε, ζητήσαμε κάτι που δεν έχει συμπεριληφθεί στον τελικό κατάλογο ψηφοφορίας να ψηφίσουμε την 74 που είναι κοινή ΕΛΚΑ και Σοσιαλιστών. Ε, να την ψηφίσουμε πριν την 6 της Ήτρε, γιατί φαίνεται ότι φέρουν επί του ιδίου αντικειμένου αυτές οι δύο τροπολογίες για την ε, συλλογική επανόρθωση, collective redress και καλό είναι να ψηφίσουμε τροπολογία 74 γιατί θα τύχει η μεγαλύτερη συνένεση και στη συνέχεια θα καταπέσει η έξι τη Ήτρε. Πρόεδρος, ναι, ναι, το λέει εδώ. Ε, μα, α, ε, Σοφή, ε, συγγνώμη, δημιουργήθηκε σύγχυση για δεν ήξερα αν είχε προταθεί η έξι Ωραία, αποσύρω το έτοιμά μου. Να έχουμε πολλά έξι γιατί την, ε, αυτή είναι η έξι της Ήτρε. Και μετά θα κάνουμε ακριβώ αυτό που είπατε με την 6 τη ΙΜΚΟ. Ήτρε 6 λοιπόν, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήτρε 2. Υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Ήμκο 6 καταπίπτει τώρα. 75 το υπέρ, κατά. Πάλι παρακαλώ, ε, ψηφίστε πάλι για την 75 υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 76. Καταπίπτει. 77. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 77. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Τι γίνεται, γιατί σηκώνετε τα χέρια εκεί πίσω, δεν κατάλαβα. Συμβαστική F. Δύο τμήματα. Το πρώτο το κομμάτι είναι χωρίς ε, τη φράση as the sole instrument και το inability to pay. Α, όχι, αφαιρείται ολόκληρο το κείμενο, λέει η πρόεδρος, ναι. Γιατί είναι με παχιά γράμματα τότε το inability to pay και το sole instrument. Λοιπόν, βγάζουμε από το πρώτο τμήμα, από το concerned μέχρι το end. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Ναι, εγκρίνεται. Τμήμα 2. Συμπεριλαμβάνεται αυτή η παράγραφος, έτσι. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος παρακαλώ. Για το τμήμα 2 της συμβαστικής F. Πέρας. Εγκρίνεται. Εγκρίθηκαν και τα δύο τμήματα, λέει η Πρόεδρος. Ε, λοιπόν, τμηματική ψηφοφορία. Α, μέχρι τον dominant position, υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 83, highlights και μετά, υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 84 αποσύρεται, 85 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 85 παρακαλώ. Ψηφίστε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια. Παράγραφος 21 πρωτότυπο υπερκατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 89 έχει και προφορική τροπολογία του ΕΛΚ. Εδώ υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Να 90 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 8 υπέρ, κατά, Δεν είδα, δεν πρόλαβα το ΕΛΚ. Α, είστε υπέρ. Πολύ ωραία. Αποχές, άρα εγκρίθηκε. Ήμκο 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ίμκο 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 93 ε, σε δύο τμήματα. Το πρώτο κομμάτι από το expects μέχρι το sector υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα από το failing that μέχρι το form υπέρ. Κατά Αποχές. Νομίζω εγκρίνεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το πρωτότυπο για την 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 95 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 95 παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. 96 υπέρ. Ζητώ συγγνώμη, λέει η Πρόεδρος. Το πρωτότυπο της παραγράφου 27 πρώτα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα η 96 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 100 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πρωτότυπο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 99 υπέρ Πρώτο τμήμα, underlines και τα λοιπά υπέρ. Κατά αποχές, ε, ηλεκτρονικός έλεγχος. Voted. Πέρας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Calls upon investigation υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική G, υπέρ. Ε, αποφασίστε τι θα ψηφίσετε. Υπέρ. Κατά τώρα. Αποχές. Έλεγχος παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι πέρας. Εγκρίθηκε. 105 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. ΙΜΚΟ 7, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 7, σε δύο τμήματα. Το πρώτο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 8, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 11 έχει και προφορική τροπολογία και είναι και σε τρία τμήματα. Ε, γίνεται δεκτή η προφορική τροπολογία. Λοιπόν υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, ε, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα, request μέχρι το purpose υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ, κατά ε, αποχές απορρίπτεται. 106 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα, χωρίς το εδάφιο που λέει του clarify και τα λοιπά. Όλα εκτός από αυτό, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται και μετά με αυτό το εδάφιο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική εφεγκρίθηκε Ένα λεπτάκι να δω για να δούμε αν θα ψηφίσουμε την 107. Ξαφανίστηκε. Α, ναι. Εγκρίθηκε κατά πίπτη 107 λοιπόν. Το πρωτότυπο τώρα για την ε, παράγραφο 31 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται 108 υπέρ ε, κατά αποχές απορρίπτεται ε, το πρωτότυπο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Citations 1 έως 20 ομαδών υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 Κατά ε, αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 4 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, η 5 ε, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 8 ε, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 9 είπε σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, whereas και τα λοιπά, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, whereas μέχρι τις startups, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. δέκα υπέρ κατά. Ένα λεπτάκι. Μην τα... Για να είμαστε σίγουροι έλεγχος, παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Μάλιστα εγκρίθηκε. Ε, συμβαστική H. Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Η 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Και τώρα ψηφίζουμε το τροποποιημένο κείμενο. Ηλεκτρονικός ε, θα... Ε, συγγνώμη, ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Παρακαλώ. Πέρας. 33 ψήφοι υπέρ, κανείς κατά, 6 αποχές. Συγχαρητήρια για τον εισηγητή μας. Ωραία. Τώρα ε, περνάμε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είσαστε έτοιμοι. Ε, λυπάμαι, λυπάμαι που μας παίρνει τόσο πολύ χρόνο, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Παράγραφος 1, αρχικό κείμενο, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 2, 7, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 8, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 9, προφορική τροπολογία και δύο ξεχωριστά τμήματα. Ε, είναι μια προφορική τροπολογία των σοσιαλιστών και δημοκρατών. Ψηφίζουμε λοιπόν το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τμήμα 2 υπέρ, κατά, αποχές ε, απορρίπτεται. Η 10 αποσύρεται, 11 υπέρ, κατά, αποχές Θέλετε να ελέγξουμε την 11. Ελέγχουμε την 11. Πέρας. Απορρίπτεται όπως βλέπετε. Αρχικό κείμενο της παραγράφου 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται άμα θέλετε ας ελέγξουμε. Αλλά τη στιγμή που συντηρητική και το ΕΛΚ μαζί υπάρχει πλειοψηφία. Λοιπόν, ψηφίζουμε, μπάση περιπτώσει, την 12. 12. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεκατρία προφορική του ΕΛΚ. Την έχετε όλοι, την προφορική, τη 13. Ευχαριστώ. Θα θέλαμε να προσθέσουμε τη λέξη more στην ε, προφορική της Ευαζολή, δηλαδή τη λέξη more πριν από το transparent. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο, παράγραφος 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε την 15. Ελέγχουμε λοιπόν την 15. Ε, ανοίγει η ψηφοφορία, αρχίζει, ψηφίσατε όλοι, πέρας και όπως βλέπετε απορρίπτεται. Λυπάμαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Συμβιβασμός χωρίς αριθμό που καλύπτει τις 17-18, 16-17-8 17 18 κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Ένα. Η ένα έχει αποσύρθει καθώς και 2 και 3, 4 υπέρ, υπέρ της 4 κατά αποχές απορρίπτεται, 5 αποσύρεται, 6 με μία προφορική, αντί 30% έχουμε 23% υπέρ, κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το κείμενο όπως έχει τροποποιηθεί υπέρ. Κατά. Είσαστε κατά. Ας γίνει, ας το κάνουμε με τις κάρτες μας. Λοιπόν, τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική. Αρχίζει. Πέρας. 37 υπέρ, 4 αποχές. Παρά ορισμένες αλλαγές, τώρα ψηφίζουμε την ε, εφαρμογή του ΕΝΟΕΙ χώρου πληρωμών σε ευρώ. ΣΕΠΑ, παράγραφος 1. Τροπολογία της Αρλίν Μακάρθη υπέρ, κατά, αποχές ε, θεωρώ ότι εγκρίνεται. Παράγραφος 2. Ε, Άλλην Μακάρθι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε στο κείμενο όπως έχει τροποποιηθεί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ωραία. Γρήγορα πάμε. Θαύμα. Αυτό ήταν, αυτή ήταν η προφορική. Τώρα φτάνουμε στο ψήφισμα. Παράγραφος 1. Αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 2. Τροπολογία σοσιαλιστών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 3. Αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 4. Σοσιαλιστές υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αποσύρονται οι επόλοιπες. Αρχικό κείμενο της παραγράφου 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άλλη Μακάρθη 4 νέο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η επόμενη αποσύρεται. SND της παραγράφου 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. σοσιαλιστές, ε, τροπολογία της 6, αντί economical economic. Κάποιος ζήτησε το λόγο. Ναι, δεν ξέρω αν ε, συμπεριλαμβάνεται αυτό σε όλους τους κατάλογους πληροφορία, αλλά θα ήθελα να προσθέσουμε, αν συμφωνούν οι συνάδελφοι, το εξή στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη σειρά όπου αναφέρεται respective consultation, να πούμε including all stakeholders, να συμπεριληφθούν δηλαδή όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς. Είναι αυτονόητο, αλλά για λόγους πληρότητες. Και από το τέλος η πέμπτη σειρά μεταξύ το banking sector και το commission θα πρέπει να αναφέρεται payment sector κανονικά. Όχι banking sector, payment sector. Λοιπόν, θα θέλαμε να διορθωθεί αυτό αν συμφωνούν οι συνάδελφοι. Ωραία, λέει η πρόεδρος υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο, παράγραφος 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Σοσιαλιστές, παράγραφο 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα έχουμε την ε, τροπολογία της 8α υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προήμια 1 έως 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Προήμιο α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΒΑ καινούριο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σοσιαλιστές στο ΣΥ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία συμβασμού Α υπέρ κατά Δεν υπάρχει ξεχωριστή ψηφοφορία, δεν τη βλέπω τουλάχιστον εγώ. βλέπω επικρατή σύγχυση. Νομίζω ότι όλο το κείμενο έχει αντικατασταθεί με το κείμενο που βλέπετε. Συμφωνείτε υπέρ του α κατά αποχές εγκρίνεται. Έχοντας υπόψη δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σίγμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, I υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, J α υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται κάπα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα θα δούμε το σύνολο της τροπολογίας όπως έχει τροποποιηθεί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Νομίζω ότι θα πρέπει να ψηφίζουμε σε μπλοκ όπου μπορούμε συνάδελφοι. Λοιπόν, τώρα τελειώσαμε με τον ενιαίο χώρο και έχουμε τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Πώς θα καταστούν αποτελεσματικές. Έχουμε μία, έχουμε μία ενιαία ψηφοφορία. Ποια είναι υπέρ του προσχεδίου, μάλλον της προφορικής ερώτησης. Α, είναι καταρχήν η προφορική σας ερώτηση, η υπέρ της προφορικής κατά αποχές εγκρίνεται. Και στη συνέχεια έχουμε τι έχουμε, έχουμε και πρόταση ψηφίσματος. Ωραία, πρόταση ψηφίσματος, παράγραφος 5α, νέα, υπέρ, κατά, Θα ελέγξουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Άρα, η ξεχωριστή ψηφοφορία στο κείμενο συμβιβασμού δεν κατανοώ τι πρέπει να γίνει. Ο συνήθως. What? Ψηφίζουμε ξεχωριστά στο κείμενο συμβασμού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε στην πρόταση όπως έχει τροποποιηθεί υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Ωραία. Πέρας ψυχοχωριών. Τώρα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων με, λέει η πρόεδρος και διακόπτη, με τον κύριο Ακερχόλμ, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλευτικού Φορέα για την διακυβέρνηση στον τομέα της στατιστικής. And you have had the first report. Και νομίζω ότι θα έχετε λάβει την πρώτη ετήσια έκθεση. Um, Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα έχουμε μία ανταλλαγή απόψε με τον κύριο Άκερχολμ, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλευτικού Φορέα. Χάσαμε χρόνο λόγω ψηφοφορίας. Ο κύριος Άκερχολμ θα, κάνει, θα μας κάνει μία σύντομη εισήγηση 5 7 λεπτών και μετά θα αρχίσει η συζήτηση. Σα Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και για την ε, πρόσκληση για να σας παρουσιάσω κάποιες θέσεις για πολύ βασικά θέματα. Το Μάρτιο του περσινού έτου υποτίθεται ότι θα ξεκινήσαμε τις εργασίες μας και θα θέλαμε να προετοιμάσουμε μια έκθεση για το φθινόπωρο. Δεν έχουμε λοιπόν πολύ χρόνο και γι' αυτό αναγκαστήκαμε να επικεντρωθούμε σε τρία θέματα. Uh, Στην επαγγελματική ανεξαρτησία που ασφαλώς αποτελεί και τον πυρήνα. Το δεύτερο θέμα ήταν οι πόροι που αν ήδη αποτελεί πρόβλημα το θέμα αυτό, πρόκειται να αποτελέσει ακόμα πιο πολύ μεγάλο πιο πρόβλημα στο μέλλον. Και το, τρίτο θέμα ήταν η δέσμευσή μας στην ποιότητα. Αυτό λοιπόν που κάναμε είναι το, το εξή. Αναγκαστήκαμε να στριχθούμε στις ε, διατηθέμενες πληροφορίες βάσει των εκθέσεων αξιολόγησης και διοργανώθηκαν και ακροάσεις με διάφορα μέρη για να εκτιμηθεί η συνεργασία στον στατιστικό τομέα εντός του εσωτερικού της Ένωσης. Εν γέννη, φαίνεται ότι σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά η πρόοδος αυτή περιορίζεται πιο πολύ στον προγραμματισμό και όχι τόσο πολύ στην εφαρμογή. Και άρα ένα από τα γενικά μηνύματα που θέλουμε να αποστείλουμε είναι ότι χρειαζόμαστε πιο πολύ εφαρμογή, πιο πολύ υλοποίηση σε ό,τι αφορά την επαγγελματική ανεξαρτησία. Έχει σημειωθεί κάποιες, ε, κάποια πρόοδο στην νομική υποστήριξη και κάποια πρόεδρος, πρόοδος συγγνώμη, για να ε, εξασφαλίσουμε την πρακτική εφαρμογή. Υπάρχουν κάποια θέματα στα οποία θα πρέπει να δώσουμε προσοχή μια υποψία παρέμβασης η οποία θα επηρέαζε ενδεχομένως την ποιότητα των στοιχείων και πολλά θέματα διορισμού και απόλυσης των ε, επικεφαλής των ε, στατιστικών υπηρεσιών. Η Eurostat από αυτή την άποψη αποτελεί έναν ιδιαίτερο οργανισμό γιατί αποτελεί εκ παραλλήλου και γενική διεύθυνση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ αποτελεί ανεξάρτητη αρχή στατιστικών στοιχείων της Ένωσης. Άρα θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η επικοινωνία και το έργο της δεν θα θεωρείται μόνο ανεξάρτητο, αλλά και θα είναι ανεξάρτητο. Σε αυτό και αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το τμήμα της επικοινωνίας. Και η Επιτροπή πάντα, τα άτομα της Επιτροπής μιλούν πάντα εξ ονόματος της Επιτροπής. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο θέμα, τους πόρους, να επιστήσουμε την προσοχή στο ότι θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη θέση προτεραιοτήτων, καλύτερη συνεργασία στο ιστορικό της Ένωσης, να χρησιμοποιούνται καλύτερα οι βέλτιστες πρακτικές προκειμένου να εξοικονομηθεί κόστος. Επίσης, να εξετάσουμε ποια είναι η συνεργασία ανάπτυξης που μπορεί να επιτευχθεί για τη μείωση του κόστους. Επίσης, τονίζουμε την ανάγκη διασφάλισης ε, σωστών εκπαιδευτικών συστημάτων προκειμένου να προσελκύσουμε τους πιο καλούς στατιστικολόγους. Επίσης, να τονίσουμε ότι οι μεγάλες διακυμάνσεις στους οικονομικούς πόρους θα μπορούσαν να αποβούν επιζημίες για τη στατιστική παραγωγή μακροπρόθεσμα σε ό,τι αφορά τη δέσμευση για την ποιότητα. Σημειώνουμε ότι πολλά έχουν γίνει εντός του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος σε ό,τι αφορά τις νέες διαστάσεις και δραστηριότητες ποιότητες και τις ε, νέες κατευθυντήρες οδηγίες, αλλά χρειαζόμαστε την ε, ισχυρή δέσμευση των μεγάλων διευθυντικών στελεχών, προκειμένου να σημειωθεί όντως πρόοδος. Σε ό,τι αφορά τον συντονισμό, υπήρξε μεγαλύτερο συντονιστικός ρόλος όντως για τη Eurostat και να τονίσουμε ότι αυτό θα πρέπει να γίνει απόλυτα σεβαστό, ιδιαίτερα στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των στατιστικών στοιχείων και να μην είναι υπερβολικά μεγάλο και το βάρος της συλλογή των στατιστικών στοιχείων. Το ίδιο φυσικά ισχύει και σε εθνικό επίπεδο. Ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών δυστυχώς δεν επέλεξαν να τηρήσουν τον κώδικα αυτό παρά το γεγονός ότι η παραγωγή στον κλάδο αυτό λίγο πολύ ακολουθούν τους ίδιους κανόνες. Τονίσαμε επίσης την ανάγκη για μεγαλύτερο συντονισμό, συνεργασία και απονομή ευθυνών στο, μεταξύ ε, των Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών και της Eurostat. Τέλος, η Επιτροπή για την εποπτεία των χρηματοοικονομικών και των ισολογισμών δραστηριοτήτων θα πρέπει να συνεχίσει τις αλλαγές που έχει ξεκινήσει. Τις μεταρρυθμίσεις που έχει ξεκινήσει. Όταν ολοκληρώσαμε λοιπόν τη διαδικασία αυτή και ήμασταν στη φάση δημοσιοποίησης της, ε, των στοιχείων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέκυψε η περίπτωση της Ελλάδας, η υπόθεση της Ελλάδας. Και αυτό φυσικά έχει να κάνει και με την ΕΣΚΑΠ, γιατί αυτή ξεκίνησε βάσει των εμπειριών της 2004 και 2005 τις ε, διαδικασίες αυτές. Όπως ε, όταν λοιπόν ξεκίνησε η διαδικασία αυτή, είχαμε μόνο κατακαιρματισμένες πληροφορίες στην διάθεσή μας. Δεν είχαμε τη δυνατότητα, δεν είχε τη δυνατότητα η ΕΣΚΑΠ να αντιδράσει. Και δεν είχε χρόνο ουσιαστικά να αφιερώσει στην έκθεση την πλήρη έκταση στο θέμα αυτό. Σήμερα ανακύπτει λοιπόν μια νέα κατάσταση, την οποία ακόμα δεν έχουμε αναλύσει πλήρως. Ωστόσο, θεωρούμε ότι δύο είναι τα συμπεράσματα τα οποία ήδη διαφαίνονται στην παρούσα φάση. Το πρώτο είναι το εξή. Είναι σαφές ότι μπορεί να υπάρχουν υποθέσεις όπου χρειάζεται ε, καλύτερη παρακολούθηση των μεθόδων και των ε, πρακτικών που εφαρμόζονται σε κάθε χώρα σε σχέση με το τι προβλέπεται σήμερα. Και γι' αυτό λοιπόν η ΕΣΚΑ προτείνει να δοθούν πιο πολλές αρμοδιότητες εποπτείας στη στάτ. Αλλά αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Καταρχάς ότι θα πρέπει να είναι σαφείς οι βασικοί κανόνες για την εφαρμογή και κατά δεύτερον ότι τέτοιες διατάξεις θα πρέπει να υποστηρίζονται από τους απαραίτητους φόρους προκειμένου να είναι αξιόπιστες. Κάτι άλλο. Η ίδια η ΕΣΚΑΠ ότι η ΕΣΚΑΠ θα πρέπει να μας δίνει τα απαραίτητα μέσα για να μπορέσουμε να εγγυόμαστε τη σωστή εφαρμογή του κώδικα στην σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό φυσικά το προγραμματίζουμε σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη τους πόρους που έχουμε φυσικά και στη διάθεσή μας. Επίσης, να τονίσω ότι στην επόμενη έκθεση την οποία ξεκινήσαμε να καταρτίζουμε, θα συνεχίσουμε να εστιαζόμαστε στα τρία βασικά θέματα του κώδικα, τα οποία μας απασχόλησαν και στην ε, πρώτη έκθεση. Ανεξαρτησία, ποιότητα, πόρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και εγώ. Η κυρία Ντάτη ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ. Αγαπητή Πρόεδρε, η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας μας ανησύχησε ιδιαίτερα όλους. Αναρωτιόμαστε πώς μια ευρωπαϊκή χώρα στην Ευρωζώνη έφτασε σε αυτή την κατάσταση. Όταν ανέλαβε η νέα ελληνική κυβέρνηση, τα στοιχεία του 2009 άλλαξαν από 12,7, μάλλον είχε δοθεί το στοιχείο 5,7, ενώ το πραγματικό έλλειμμα της Ελλάδας ήταν 12,7. Και γι' αυτό αυτό ε, γνωρίσαμε κλειδονισμού στην Ευρωζώνη. Υπάρχει μεγάλη ελεξάρτηση πλέον μεταξύ κρατών μελών της Ευρωζώνης. Γι' αυτό, όπως υπενθύμησε η Επιτροπή και το Συμβούλιο, θα πρέπει να συντονιστούμε, να συντονίσουμε τις οικονομικές μας πολιτικές. Ε, δεν θέλουμε να στυλιτεύσουμε την Ελλάδα, αλλά αναρωτιόμαστε πώς φτάσαμε εκεί και γι' αυτό θα θέλαμε να φτάσουμε σε μόνιμες λύσεις για να μην ξαναβρεθούμε σε αυτή την κατάσταση. Όπως είπατε και εσείς, σήμερα θα πρέπει να έχουμε αξιόλογα, μάλλον ε, σωστά στατιστικά στοιχεία. Κυρία ε, Ντάτη, μιλάτε πολύ γρήγορα. Είναι γεγονός ότι θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε εγγυημένα στατιστικά στοιχεία και είμαι πεπισμένη ότι έτσι θα μπορέσει να οδηγηθεί σε ευημερία η Ευρωζώνη. Τα ελληνικά στατιστικά στοιχεία δυστυχώς δεν ήταν σωστά και το 2005 η Ελλάδα δημιούργησε την, ε, μια ιδιαίτερη λογιστική, τη δημιουργική λογιστική, Γι' αυτό θα πρέπει να προωθήσουμε έναν κώδικα δεοντολογίας. Γι' αυτό ακριβώς η Επιτροπή στις 15 Φεβρουαρίου πέρσι όρισε έναν νέο κώδικα συμπεριφοράς και δεοντολογίας μέσα στα πλαίσια το, της, αξιό, της αξιολόγησης των στατιστικών στοιχείων. Πιστεύετε λοιπόν ότι ε, δεν υπάρχει δυνατότητα πλέον παραχάραξης των στατιστικών στοιχείων. Τι προτείνετε έτσι ώστε να θέσουμε τέλος σε μια παρόμοια κατάσταση. Η δική σας Επιτροπή δεν θα πρέπει να έχει νέες αρμοδιότητες έτσι ώστε να μπορέσει να προωθήσει αυτή την εποπτική διαδικασία. Πρόεδρος, πολλά μέλη θέλουν το λόγο. Επειδή έχουμε πολύ περιορισμένο χρόνο, ίσως θα ήταν σκόπιμο να υποβάλουμε ερωτήσεις όλοι και να συγκεφαλαιώσετε στο τέλος. Ο Ζαν Πολ. Θα είμαι σύντομος, ε, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή σας υπάρχει εδώ και λίγο χρόνο, άρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ανεπάρκεια εργασίας. Θα ήθελα να σας ε, ρωτήσω ε, κατά πόσο δεν είστε αφελείς, διότι σήμερα στυλιτεύουμε στην Ελλάδα σαν να ήταν η μόνη. από το 2000 όμως παραχαράσσονται τα στατιστικά στοιχεία Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη σύγκρουση συμφερόντων και άρα ε, υπάρχει μεγάλη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ υπαλλήλων της Eurostat και αξιωματούχων των κρατών μελών ή ορισμένων τραπεζών. Και μέσα στα πλαίσια αυτή της σύγκρουσης θα πρέπει να δούμε τι στοιχεία προωθούνται. Μιλάμε ήδη για στοιχεία του 2000. Όταν ένας υπάλληλο τη ε, ε, Eurostat είχε τόσες πολλές προσφορές από τράπεζες, ε, στην ουσία έπρεπε να βρει μια σολομόντιο λύση. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι πολλά στοιχεία είναι ήδη απαρχαιωμένα Υπάρχουν, ε, υπάρχει μεγάλο δέλεαρ προς τους ευρωϊπαλλήλους, γι' αυτό δεν θα πρέπει να είμαστε καθόλου αφελείς. Ε, δεν, υπάρχει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην προσπαθήσουν πολλοί να χρηματίσουν τους ευρωϊπαλλήλους. Ο Ούντο. Ελαμβάνοντα υπόψη την οικονομική κατάσταση των κρατών μελών, την χρηματοοικονομική τους κατάσταση, θα ήθελα να υποβάλω δύο, τρία μπλοκ ερωτήσεων. Καταρχήν, οι κερδοσκόποι προβαίνουν σε έναν αγώνα δρόμου, όπου αφήνουν και πολλά θύματα από την χρηματοπιστωτική αυτή κρίση. Δεν μας αφορά αυτό, διότι εσείς τουλάχιστον δεν είσαστε αρμόδιος επί του θέματος. Το λέω απλώς διότι στυλιτεύουμε ορισμένα μεμονωμένα κράτη σαν να έφεραν όλο το βάρος της κατάστασης, κάτι το οποίο δεν ισχύει. Δεύτερο σημείο. Και εδώ προσεγγίζουμε την ΕΣΚΑΠΑ. Θα είμαι λιγότερο ευγενικό από ότι ο Υπάρχουν ιδιωτικέ τράπεζε οι οποίε ε, συμβουλεύουν τα κρατή-μέλη για, την, ε, ε, για τα στοιχεία του, τα στατιστικά του στοιχεία και υπάρχουν προβλήματα σε ό,τι αφορά την εκτίμηση της κατάστασης των δεδομένων και τα κράτη-μέλη αρνήθηκαν πριν από κάποιο καιρό να δώσουν περισσότερες αρμοδιότητες στην Eurostat. Θεωρείτε ότι λόγω της τρέχουσας κατάστασης θα υπάρξει κάποια αλλαγή στην, ε, σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες της Eurostat, προκειμένου να συμπεριληφθούν και τα κεντρικά αυτά τα δεδομένα. Το τρίτο πρόβλημα όμως είναι ένα πρόβλημα ουσίας. Και αυτό ισχύει όχι για ένα, αλλά για περισσότερα κράτη-μέλη. Έχετε την εντύπωση ότι η τα δεδομένα βάση στα κάθε, στο κάθε, κάθε κρατός μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τα δημόσια, τις δημόσιες υπηρεσίες και σε ό,τι αφορά και τις ιδιωτικές εταιρείες είναι σωστά. Δηλαδή τελικά τα ομαδοποιημένα δεδομένα είναι αληθή Γιατί αν δεν είναι σωστά αυτά τα μεμονωμένα στοιχεία, πώς είναι σωστά αυτό, πώς μπορεί να είναι σωστά τα ομαδοποιημένα κεντρικά στοιχεία, τα κεντρικά δεδομένα. Τι σημαίνουν δηλαδή αυτά τα ομαδοποιημένα κεντρικά δεδομένα. Δεν θα πρέπει να υπάρχει κάποιο κεντρικό σύστημα το οποίο θα εξασφαλίζει ότι γίνεται σωστή συλλογή των βασικών αυτών δεδομένων. Ο κύριος Κλέντς, ευχαριστώ. Για τα θέματα αρμοδιότητας τα έχουμε δείξει ήδη. Δεν θα επεκταθώ. Σε πολλούς τομείς που είναι πολύ κρίσιμοι προσπαθούμε να ε, καταρτήσουμε σωστούς μηχανισμούς ε, πρόληψης σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τη μηχανική κατασκοπία, σε ό,τι αφορά την απάτη, την διαφθορά. Η Eurostat έχει έναν ιστορικό τομέα ο οποίος ε, καταβάλει προσπάθειες βάσει συγκεκριμένων ενδείξεων να εντοπίσει περιπτώσεις ε, απάτης ή τουλάχιστον ε, τέτοιους μηχανισμούς περίεργους. Κατά δεύτερον, γίνονται σφάλματα κατά κανόνα από τους υπαλλήλους. Οι υπάλληλοι είναι και αυτοί οι μέλη των 27 κρατών μελών. Άρα υπάρχει και η υποψία τουλάχιστον ότι ένας Έλληνας υπάλληλο, για παράδειγμα, στην περίπτωση της Ελλάδας θα είναι πιο προσεκτικός από ότι κάποιος άλλος, άλλης εθνικότητας. Πώς λοιπόν διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει τέτοια σύγκρουση συμφερόντων λόγω της εθνικότητας των υπαλλήλων. Um, σας ευχαριστώ, Έντουαρτ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Άκροχολμ, είμαι βέβαιος ότι έχετε πολύ μεγάλη δουλειά μπροστά σας και καταλαβαίνουμε φυσικά ότι δεν είναι όλα τα στατιστικά στοιχεία το ίδιο. Άλλο να μετράμε τα πουλιά που περνάνε πάνω από μια χώρα και άλλο να μετράμε το ΑΕΠ και τα δημοσιονομικά γιατί φυσικά εδώ πέρα υπάρχουν και άλλοι σκοποί και αναφέρομαι στα πρότυπα της Ευρωζώνης και του καθεξής. Το θέμα της ε, διοργάνωσης επισκέψεων και συνομιλιών με τα άτομα αυτά στις ε, υπηρεσίες στατιστικής είναι σημαντικό. Αλλά όταν τίθεται θέμα απάτης, θα πρέπει να εξαρτώμαστε από τα άτομα επιτόπου. Γιατί ξέρω από την εμπειρία μου ότι το θέμα είναι να έρθει μια αντιπροσωπεία να μιλήσει με το προσωπικό να φύγει Όλα αυτά είναι χρήσιμα, αλλά θα πρέπει να στηριζόμαστε στους υπαλλήλου επιτόπου. Αυτοί μπορούν να μυριστούν πραγματικά αν υπάρχει πρόβλημα με τα δεδομένα ή όχι. Και τέλος, να πούμε ότι πολλές φορές τα δεδομένα αναφέρονται ότι είναι αληθή ή όχι, αλλά η πηγή, τα πρότυπα λογιστικής των δημοσιονομικών είναι τόσο παροχημένα και ξέρω περιπτώσει βασίζονται για παράδειγμα στι χρηματικέ ροέ, Δεν βασίζονται δηλαδή σε σωστέ αρχέ. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω την άποψή σα σχετικά. Um, σας ευχαριστώ πολύ. κανεί άλλος παρακαλώ. Να δώσω και κάποιο ιστορικό υπόβαθρο, γιατί ήμουν εισηγήτρια για την σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλευτικού Φορέα. Και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων από πλευρά Κοινοβουλίου προσπαθήσαμε να σας δώσουμε πιο πολλές αρμοδιότητες. Και είχαμε την τη Προεδρία τον κύριο Ανταμάκ από την άλλη πλευρά. Νομίζω όμως ότι τα κράτη-μέλη δεν ήθελαν ήταν σαφές ότι δεν ήθελαν να δώσουν πιο πολλές εξουσίες σε ό,τι αφορά την ε, διερεύνηση των στατιστικών τους δεδομένων και τελικά δεν πέτυχε το Κοινοβούλιο όλα όσα ήθελε. Τώρα λοιπόν και από πλευρά Κοινοβουλίου εξετάζουμε με μάλλον ε, διστακτικό τρόπο αυτή την κατανομή των ε, αρμοδιοτήτων όπως θεωρείται θα πρέπει να γίνει το Συμβούλιο. Δεν εντάσσονται στις στατιστικές ε, ε, στο δυτικό κλάδο το οποίο θα τα έκανε να υπάγονται αυτόματα στη απόφαση. Το Κοινοβούλιο θα είναι στην πλευρά σας, θα σας υποστηρίξει φαντάζομαι για την αναζήτηση περισσότερων εξουσιών. Υπάρχει και το πάνελ φυσικά το οποίο δημιουργήθηκε παράλληλα για τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να υπάρχει και input, να δίνονται στοιχεία σχετικά με την ορθότητα των ε, στατιστικών δεδομένων που συλλέγονται. Αυτά λοιπόν ήθελα να αναφέρω στην παρούσα φάση. Δεν είναι κάποια ερώτηση, ουσιαστικά θα σας θέτω κάποια ερώτηση, αλλά ήθελα απλά να δώσω περισσότερες πληροφορίες. Αν θα θέλετε να μας απαντήσετε τώρα, έχουμε 10, 12 λεπτά στη διάθεσή μας. Μάλιστα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις, όχι απαραίτητα με την ίδια σειρά, όπως τέθησαν οι ερωτήσεις δηλαδή. Πρώτον, περί ε, αφέλειας. Ελπίζω ότι δεν επικρατεί αφέλεια μετά από όλα αυτά που βιώσαμε, δεν θα έπρεπε. Και επίσης, ε, καλό είναι να μην ε, στυλιτεύουμε κάποιες συγκεκριμένες χώρες, γιατί σε οποιονδήποτε θα μπορούσε να συμβεί. Και ένα σύστημα χρειαζόμαστε για να εντοπίσουμε τον κίνδυνο το νωρίτερο δυνατόν αν υπάρχει σαφώς απάτη, ε, η θελημένη απάτη, ξέρετε είναι δύσκολο να εντοπιστεί. Θα κάνουμε αυτό που μπορούμε. Το πρόβλημα, η πρόκληση με το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα είναι ότι όλα τα βασικά δεδομένα συλλέγονται σε εθνικό επίπεδο και μετά τα επεξεργάζεται η Eurostat. Η Eurostat δεν μπορεί να αναβαθμίσει την ποιότητα. Είναι κακή η ποιότητα των αρχικών δεδομένων. Κακά θα παραμείνουν τα δεδομένα μετά την επεξεργασία της Eurostat. Δεν μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα η Eurostat. Ε, και για την ποιότητα και για την αξιοπιστία σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να δράσουμε. Σε επίπεδο της πηγής. Κάτι άλλο που περιέπλεξε πάρα πολύ το θέμα των εθνικών λογαριασμών είναι η δημιουργική λογιστική που γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια. Όταν λέμε ότι οι τραπεζίτες ε, απασχολούν ε, ανθρώπους που γνωρίζουν τα περιστατιστικών δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μια στατική κατάσταση και δεν γίνονται όλα κακοί την ε, Υπάρχουν πολλοί που χρειάζονται τις πληροφορίες για να κατανοήσουν ακριβώς ε, πώς καταγράφονται διάφορες συναλλαγές στο στατιστικό σύστημα. Καλόβουλες προσπάθειες δηλαδή. Τι θα πρέπει να κάνουμε, να μετεξελίξουμε το σύστημα, να προάγουμε τη διαφάνεια, ούτως ώστε οι πληροφορίες αυτές να μην έχουν τόσο μεγάλη αξία στην αγορά. Ε, αυτό θα γίνει ενισχύοντας τη διαφάνεια στο βαθμό του δυνατού και ε, να, ε, πρέπει να επιδιώξουμε την διαθεσιμότητα των πληροφοριών με ομοιόμορφους κανόνες και ομοιόμορφες μεθοδολογίες για την καταγραφή των οικονομικών συναλλαγών. Κάτι άλλο τώρα, μας δείχνει η εμπειρία, ή τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ, η ΕΣΚΑΠ πρέπει να υπομειστεί την ευθύνη της για να ελέγξει την, το όλο οικοδόμημα, να δει δηλαδή κατά πόσο το σύστημα που έχουμε δημιουργήσει μπορεί να υποστηρίξει την αξιοπιστία του συστήματος. Υπάρχουν ε, επιπρόσθετοι έλεγχοι, έχουμε ανεξάρτητους ελεγκτές που με πάση ελευθερία μπορούν να δώσουν την αξιολόγησή τους χρησιμοποιώντας τις επαγγελματικές γνώσεις και μόνο και καμία εξωτερική επιρροή. Τώρα όταν μιλάμε για την ε, εφαρμογή ε, δεν δεν έχουμε τους απαιτούμενους πόρους για να το ελέγξουμε εμείς αυτό. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και τελικά αυτό θα παραμείνει ε, στο θέμα της ε, Eurostat. Η Eurostat πρέπει να έχει πόρους, μεθοδολογίες και δυνατότητες ούτως ώστε να εντρυφεί επαρκώς στο σύστημα για να διεξαγάγει και τους απαιτούμενους ελέγχους μεριμνώντας ώστε οι πληροφορίες που λαμβάνει προς συνάρθρηση να είναι επαρκείς και ακριβείς. Η νομοθεσία δεν ε, ε, εκχωρεί αρκετή αρμοδιότητα στη Eurostat ώστε να σκάψει βαθύτερα στο σύστημα και να το ελέγξει. Ε, έχουν γίνει πάρα πολλές επισκέψεις, πολλές συζητήσεις. Συζητήσεις σε σχέση με την ίδια την οικοδόμηση του συστήματος και είμαι σίγουρος ότι όλα αυτά ήταν σωστά, αλλά τελικά τι προκύπτει. Οι πληροφορίε με τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκαν δεν οδηγούσαν σε σωστά αποτελέσματα. Ε, και πώς το αντιλαμβάνομαι εγώ η Eurostat δεν είχε ε, την αρμοδιότητα, την ισχύ για να προχωρήσει περισσότερο. Η ESCAP ε, θα επικουρήσει την Eurostat λοιπόν για να μπορέσει να επομιστεί αυτή τη την ευθύνη όπως είπα και στην αρχική μου παρουσίαση, χρειάζεται να έχουμε και πόρους υποστηρικτικούς. Δεν γίνεται να προβλέπετε ευθύνη, να, αλλά να μην έχουμε, δεν γίνεται να μην έχουμε τους απαιτούμενους πόρους μέσα στο σύστημα για να κάνουμε τους ελέγχους που προκύπτει ότι χρειάζονται. Άλλε αρμοδιότητες της ΕΣΚΑΠ τώρα σε αυτή τη διαδικασία, κοιτάζω και την ώρα, Ενδιαφέρον το ερώτημα, Πρόεδρε, αλλά δεν έχουμε ακριβώς ε, ε, επαρκείς πληροφορίες προς το παρόν. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα ελέγχει την κατάσταση η ΕΣΚΑΠ σε μεμονωμένα κράτη-μέλη. Από όσο ξέρω, έχω την εντύπωση ότι θα χρειαστεί αξιολόγηση μεμονωμένων κρατών, ούτως ώστε να γίνει ορθή αξιολόγηση του συνόλου του συστήματος και να καθοδηγήσουμε ορθά την λειτουργία του συστήματος. Μας δείχνει η εμπειρία ότι η νομοθεσία προβλέπει αυτή τη δυνατότητα και οι επόμενες εμπειρίες μας θα μας δείξουν αν επαρκεί αυτή η νομοθεσία. Ε, προβλέπει η νομοθεσία ότι σε δύο-τρία χρόνια θα επανέλθουμε για ενδιάμεση αξιολόγηση. Κατά πόσο ενδείκνεται η νομοθεσία που έχουμε εγκρίνει. Θα έχουμε πολύ περισσότερες εμπειρίες και θα έχουμε δοκιμάσει και τα όρια του συστήματος και θα μπορέσουμε να συμβουλεύσουμε το Κοινοβούλιο σχετικά με το αν επαρκεί το σύστημα που τώρα οικοδομούμε. Ε, τώρα, ε, για τις εσωτερικές λειτουργίες της Eurostat, Υπάρχει εκπρόσωπος εδώ της Eurostat, νομίζω ότι καλύτερα θα ήταν να απαντήσει εκείνος παρά να μιλώ εγώ εξ ονόματος της Eurostat. Πάντως, ε, κάτι σημαντικό είναι να θεσπίσουμε τα συστήματα ώστε να κάνουμε ελέγχους ε, συνέπειας ε, των διαφόρων στατιστικών στοιχείων ούτως ώστε να εντοπίζουμε ιονή προβλήματα. Ε, το θετικό με πολλά οικονομικά στατιστικά στοιχεία είναι ότι θα υπάγονται στο ίδιο σύστημα. Δηλαδή πρόκειται για διαφορετικά τμήματα του ίδιου συστήματος και αν υπάρξουν παρεκκλήσεις αργά ή γρήγορα θα αποκαλυφθεί αυτό. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε να κάνει μια σύντομη επερώτηση, ερώτηση, όχι, αλλιώς ολοκληρώνουμε, ευχαριστούμε. Ε, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το θέμα με τις